Bueno, venga, vamos a empezar Αρχίζουμε με αυτό το σημείο, λέει ο Πρόεδρος. Vamos a empezar la reunión de esta tarde porque, dada la, el gran número de diputados, cuanto Ο κόσμος ε, ψηφίζει τώρα. Όλοι είναι στην Επιτροπή Γεωργίας. Ε, είδατε που δίνουν προτεραιότητα όλοι. Πάντα τη Γεωργία και ποτέ στην ε, στην Αλία. Ε, επομένω, εδώ είμαστε, θα τα πούμε μεταξύ μα, εδώ οικογενειακά. Όσο πιο νωρί πιο νωρί θα τελειώσουμε και οπότε επομένω θα πρέπει να δούμε τι θέματα ακόμα και μα ενδιαφέρουν. Πρώτα-πρώτα έχουμε το σημείο 12 τη μεσαία διάταξη. Η πράσινη βίβλο που αφορά προκλήσει και ευκαιρίε. Προ ένα κοινό πλαίσιο στατική για τη χρηματοδότηση τη έρευνα και τη καινοτομία στην ΕΕ. Η Ήτρε είναι η κυρίως αρμοδία επιτροπή. Εμείς ζητήσαμε να γίνει σχετική έκθεση, γιατί για μας η έρευνα για την Ελία είναι θέμα κεφαλαίου σημασία. Και έχουμε άλλωστε και το τελευταίο πρόγραμμα πλαίσιο, στο οποίο με τίποτα δεν καλύφθηκαν όλα εκείνα τα οποία εμείς πάρα πάρα πολύ βάσιμα είχαμε ζητήσει. γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθεί η έρευνα για την Ελία. Επότε θα πρέπει και πάλι να κινητοποιηθούμε όσον αφορά το θέμα αυτό και αυτή τη φορά να αποσπάσουμε κάποιο αποτέλεσμα. Δεν πάση Ο αρμόδιος συνάδελφος είναι ο κύριος Βαλέσσα. Και στο όνομα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουμε τον κύριο ο οποίος ήρθε για να μας κάνετε σχετική εισήγηση. Έχετε το λόγο. Καλώς ορίσατε και η σκητάλη σε εσάς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να σας παρουσιάσω πολύ σύντομα τους προσανατολισμούς που περιέχονται στην πράσινη βίβλο της Κομισιόν για την μελλοντική χρηματοδότηση της καινοτομίας και της έρευνας. Πριν περάσω στο περιεχόμενο, επιτρέψτε μου να περιγράψω το πλαίσιο. Σύντομη εισαγωγή, αλλά θα ήθελα να κάνω μια αναδρομή. Οι επικεφαλείς κρατών και κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όταν συναντήθηκαν το Φεβρουάριο ζήτησαν από την Κομισιόν να συγκεντρώσει όλες τις σχετικές διαδικασίες και τα πακέτα σχετικά με την καινοτομία και την έρευνα στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής, ούτως ώστε να είναι πολύ πιο εύκολα προσπελάσιμη ε, προσπελάσιμο προς ενδιαφερομένους. Αυτό λοιπόν θα τεθεί σε εφαρμογή ε, το προσεχή περίοδο από το 2013. Και οι βασικές αρχές που διέπουν αυτόν τον προϋπολογισμό είναι η στήριξη των προτεραιοτήτων πολιτικής της Ευρώπης του 2020, αύξηση της προστιθέμενης αξίας και ε, μεγαλύτερη απόδοση, α, απόδοση στις δαπάνες που γίνονται. Καταρχήν, βάση είναι το υπάρχον πλαίσιο. Το πρόγραμμα πλαίσιο ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας, το γνωστό ΣΥΠ, και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που συνήθως το λέμε IT. Αυτό το στρατηγικό πλαίσιο θα προκαλέσει θεμελιώδεις αλλαγές με την δημιουργία μιας σειράς μέσων και εργαλείων, ώστε να ενισχυθεί η βασική έρευνα και η σύνδεση με την αγορά. Ταυτόχρονα προσφέρει δυνατότητες, σημαντικές δυνατότητες, ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες, να υπάρξουν τυποποιημένες ε, διαδικασίες και πρότυπα σε όλες τις φάσεις. Αρχίσαμε λοιπόν να αναπτύσσουμε τις ιδέες μας με βάση την αξιολόγηση των προγραμμάτων που ήδη τρέχουν και εντοπίστηκαν κάποιες θετικές πτυχές αλλά επίσης και κάποιες ελλείψεις και αδυναμίες. Στα θετικά τόσο το υπάρχον πρόγραμμα πλαίσιο για την ε, έρευνα, όσο και το πρόγραμμα για την καινοτομία και την τεχνολογία. Έχει βεβαίως θετικά στοιχεία, παραδείγματο χάρη τη διασυνοριακή συνεργασία και την θέσπιση μιας κρίσιμης μάζας, κάτι που καθίσταται όλο και πιο σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη το χαρακτήρα των προκλήσεων. Άρα λοιπόν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο επιτύχαμε βελτιώσεις χάρη στον ανταγωνισμό. Αυτό είναι κρίσιμη σημασία αν θέλουμε να ανταγωνιζόμαστε με πιο επιθετικό τρόπο σε παγκόσμιο επίπεδο. Τόσο το πρόγραμμα SIP όσο και το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία ε, παρουσιάζει σημαντικό ποσοστό συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αλλά επίσης και ιδιωτική χρηματοδότηση που ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία. Τώρα, στις, ε, στις ανδυναμίες. Ένα σύνθετο πεδίο δράσης και ως προς τους επιστήμονες, ε, στο πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και τεχνολογίας, ε, εντοπίζεται η ε, ανάγκη απλοποίησης των διαδικασιών. Αν θέλουμε δηλαδή να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να εστιάσουμε πιο συγκεκριμένα, πρέπει να λάβουμε υπόψη προτάσεις που λένε ότι πρέπει να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις της κοινωνίας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Και διατυπώνεται η επιθυμία ευρύτερης συμμετοχής, όπως επίσης και ανάγκη για διάκριση των θεμάτων που θέτει η κοινωνία, η κλάδοι, αλλά και οι επιστήμονες. Η πράσινη βίβλος λοιπόν έρχεται ακριβώς να καλύψει αυτές τις αδυναμίες επί τη βάση τριών στρατηγικών στόχων. Αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που έρχονται από την κοινωνία, αύξηση της ανταγωνιστικότητας και αυξάνοντας τα επίπεδα αριστείας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας. Εντοπίστηκαν λοιπόν τρία βασικά θέματα τα οποία πρέπει να καλυφθούν. Και γύρω από αυτά τα ερωτήματα ή αυτά τα θέματα η Κομισιόν προωθεί τώρα μια ευρεία συζήτηση. Τα ερωτήματα λοιπόν είναι πώς το νέο πακέτο μπορεί να οδηγήσει σε ένα ε, νέο πρόγραμμα, νέο πεδίο πιο ξεκάθαρο, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις βασικές προκλήσεις της κοινωνίας, πώς μπορούμε να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα και να έχουμε μεγαλύτερα αποτελέσματα από την προσπάθεια έρευνας και ε, από την ενίσχυση της επιστημονικής αριστείας και της έρευνας πόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να έχουμε. Έτσι λοιπόν, πράγουμε μια διαβούλευση η οποία διήρκησε τρεις μήνες και έκλεισε μόλις ε, πριν λίγες μέρες. Είχαμε τεράστια ανταπόκριση σε αυτή τη διαβούλευση. 1.300 απαντήσεις online στο ερωτηματολόγιο και περίπου 570 570 ε, έγγραφα, θέσεις και απόψεις από κυβερνήσεις, από φορείς, από πανεπιστήμια, από περιφερειακές και τοπικές οργανώσεις. Οι απαντήσεις αυτές λοιπόν τώρα αναλύονται, μόλις έφτασαν δηλαδή όπως ε, αντιλαμβάνεστε. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια προκαταρτική ανάλυση ολοκληρωμένη λίγο πριν από ένα συνέδριο που θα γίνει στις 10 Ιουνίου όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και θα διατυπωθούν κάποιες ιδέες για το πώς αυτά θα περιληφθούν σε ένα μελλοντικό πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας. Τώρα, για ενημέρωσή σας, εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν προσκληθεί για να συμμετάσχουν σε, αυτή την, σε αυτό το γεγονός, την εκδήλωση στις 10 Ιουνίου και βεβαίως επί τη βάση των ε, αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και αφού λάβουμε υπόψη την άποψη του Κοινοβουλίου και των άλλων οργάνων θα παρουσιάσουμε στη συνέχεια το πλήρες πακέτο νομοθεσίας, το πλήρες νομοθετικό πακέτο. Βέβαια είναι ακόμα πολύ νωρίς να περάσει κανείς την ανάλυση του περιεχομένου του νέου προγράμματος. Αλλά βέβαια η αλία, οι δατοκαλλιέργειες και γενικότερα τα ναυτιλιακά να είναι μέρος των προκλήσεων που προέρχονται από την κοινωνία και που θα πρέπει να ε, περιληφθούν. Πολύ σύντομα να σας πω δύο λόγια σχετικά με την έρευνα που εμείς υποστηρίζουμε στο πλαίσιο ε, του προγράμματος έρευνας και ανάπτυξης. Επτά. Στον τομέα ε, επισητισμού, τροφίμων και αλίας. Αυτή τη στιγμή υποστηρίζουμε 25 ε, προγράμματα. Το Αυτά ανέρχονται στα 70 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, άλλες... άλλα τμήματα της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης έχουμε προγράμματα για την ποιότητα των θαλασσινών και την ασφάλεια και το συνολικό πακέτο φτάνει στα 126 εκατομμύρια που ε, ουσιαστικά είναι το 15% του συνολικού προϋπολογισμού αν θέλετε σε ποσοστά. Δηλαδή πακέτο που αφορά ε, τα τρόφιμα, την βιοτεχνολογία, την ε, αλληλεία της υδατοκαλλιέργειας. 15% λοιπόν αυτού του προϋπολογισμού πηγαίνει σε αυτά τα θέματα. Επιπλέον, υπάρχει ένα άλλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. Εκεί 100 εκατομμύρια δαπανώνται για τη διαχείριση θαλασσίων οικοσυστημάτων που βεβαίως συνδέονται άμεσα με τη διαχείριση του θαλασσίου πλούτου. Έχουμε ένα άλλο τμήμα επίσης που έχει να κάνει με τις δυνατότητες, δηλαδή υποδομές και περιλαμβάνει μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Εκεί κάπου 32 εκατομμύρια ευρώ για θέματα αλίας και αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση επιλογής κάποιων άλλων προγραμμάτων στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2011. Αυτά που σας είπα ήταν του 10. Κάποιες δηλαδή δράσεις θα χρηματοδοτηθούν αργότερα φέτος από τη στιγμή που θα έχει ολοκληρωθεί η επιλογή και η ολοκλήρωση διαπραγμάτευσης των συμβολέων. Δράτω με τις ευκαιρίες για να σας επισημάνω ότι προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την τεχνολογία στον τομέα της αλίας. Έτσι λοιπόν είχαμε δύο παράλληλες δράσεις, δηλαδή ε, τρόφιμα, γεωργία, αλία, αλλά και περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές. Προσπαθήσαμε να έχουμε μια συνεκτική εικόνα με τα δύο αυτά θέματα. Ε, με τον γενικότερο τίτλο ή μάλλον κάτω από την ομπρέλα «Ο ωκεανός της αύριον». 79 εκατομμύρια διατέθηκαν για τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Αυτά λοιπόν κυρία Πρόεδρε, ασφαλώς είμαι στη διάθεσή σας να σας προσφέρω περαιτέρω πληροφορίες για συγκεκριμένες δράσεις ή να επανέλθω στην ομάδα αυτή με άλλη ευκαιρία αφού θα έχω και τα αποτελέσματα της έρευνας που έχει ολοκληρωθεί. Αν πιστεύετε ότι τούτο θα ήταν χρήσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, Dziękuję Szanowna Pani e, Przewodnicząca. E, bardzo chciałem podziękować przedstawicielowi Komisji Europejskiej za przedstawienie. Ευχαριστώ για την e, παρουσίαση αυτής της έκθεσης Βέβαια η αλληλεία και η γεωργία είναι οι βάσεις της ευρωπαϊκής οικονομίας και χρειάζονται οικονομική υποστήριξη. Υπάρχουν πολλά προβλήματα σήμερα στην αλληλεία γιατί θα πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση των πόρων του περιβάλλοντος. Επίσης ε, πρέπει να υπάρξει ολοκλήρωση των παράκτιων περιφερειών. Χρειαζόμαστε λοιπόν αποτελέσματα από έρευνες Είναι ένα μέσο αυτό το οποίο μπορεί να διασφαλίσει την θετική εξέλιξη της αλίας. Χρειάζεται όμως να πρικοδοτηθούν οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες αυτές και χαίρομαι που άκουσα θετικά πράγματα εδώ. Ε, έχουμε έτσι μια θετική τροπή σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα. Η πράσινη βίβλος όμως συγκεντρώνεται, επικεντρώνεται στην καινοτομία Τι γίνεται με την έρευνα στον τομέα της αλίας, η χρηματοδότηση της έρευνας σε αυτό το τομέα πρέπει να πάει προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. 160-150 εκατομμύρια ευρώ μας είπατε στο πρόγραμμα πλαίσιο και στο έκτο ήταν 110 εκατομμύρια. Ε, που δεν φαίνεται να χρηματοδοτείται η έρευνα της, η θαλάσσια έρευνα. Τι ακριβώς έχει γίνει, πώς καταλήξαμε σε αυτά. Στο επόμενο πρόγραμμα πλαίσιο θα αλλάξουν τα δεδομένα και πρέπει να μπορούμε να εφαρμόσουμε τους στόχους της κίνησης αλληλευτικής πολιτικής. Έχουμε μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα συζήτηση μπροστά μας και αντιπαράθεση πάνω σε αυτά τα θέματα. Θέλω να ρωτήσω όμως ε, σχετικά με τα κονδύλια εδώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν γιατί δεν τα άκουσα όλα. Τι γίνεται με την ε, υποστήριξη, τι χρειάζεται στον επιστημονικό τομέα, ούτω ώστε να γίνουν σωστές καινοτομίες και στον τομέα της αλίας. Τι νούμερα συγκεκριμένα έχετε να μας δώσετε. Ε, χρειαζόμαι περισσότερες λεπτομέρειες εδώ. Τώρα, συγκεκριμένες δαπάνες για συγκεκριμένα έργα, προγράμματα στα πλαίσια της αλίας. Σήμερα βλέπουμε μια διαφοροποίηση ενώ τώρα χρειάζονται κατεπηγόντως τέτοιου είδους έρευνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Θέλω να ρωτήσω την Επιτροπή για το πόσο ξέρουν τι έλλειμμα υπάρχει στην έρευνα για την αλία. Δεν το λέω, το λένε όλοι. Και για το ότι δεν λέγεται τίποτα το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Παλαιότερα προβλεπόταν προοικοδότησε στον προπολογισμό. Εν ώψη του 7ου προγράμματος πλαισίου, αυτό σταμάτησε. Αυτή θα πήγαινε να γίνει λογική. Και όντω το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο έχει προοικοδότηση. Όμως, η έρευνα για την αλληλεία βασικά είναι εφαρμοσμένη έρευνα. Δεν είναι το θέμα του αν θα μετράει σε ένα τα ψαράκια και δεν είναι το θέμα του κατά να δίνεται δημοσιότητα, όμως είναι απαραίτητη. Δεν το λέω εγώ, επαναλαμβάνω, το λένε όλα τα ερευνητικά ιδρύματα. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι θα πρέπει στο μέλλον να διορθώσετε τα πράγματα. Αλλιώς, λόγω του ελλείμματος στην έρευνα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Εν ώψη της μεταρρύθμισης και των δεσμεύσεων της Ευρώπης, ενώπιον του ΦΑΟ, με τα νέα οικοσυστήματα, γιατί τα οικοσυστήματα απαιτούν νέες μορφές έρευνας. Ας πούμε πολυκλαδικές. Παρακαλώ. Σκεφτείτε. Μιλήστε και με τους ανούμενες γενικές διευθύνσεις. Πώς το πρέπει να λυθεί στο μέλλον. Να διορθώσουμε τα πράγματα. Για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε το μέλλον. Είναι πολύ ενισχυτική κατάσταση. Και είναι δύσκολο προς το παρόν να διορθωθούν τα πράγματα στον προϋπολογισμό. Όλο στο τέλο δεν το λόγο. Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι, όχι, εντάξει, πρόεδρε. Αυτό που δεν μπορούσα να αναφέρω προηγουμένω είναι για το 7ο πρόγραμμα πλαίσιο το τι θα γίνει όσον αφορά αυτό που θέλουν οι επιστήμονε για να απλουστευτούν κάποιοι κανόνε, κάποιε διατάξει. Γιατί πρόκειται για κάτι το οποίο μου το είπαν πολλοί από πολλά ερευνητικά ιδρύματα. Πώς θα απλουστευτούν, θα ξεκαθαριστούν κάποιες διαδικασίες. Κάτι που οι επιστήμονες το ζητούν έντονα. Κύριε Γιώτο. Έχω, έχω μια ερωτησούλα προς την Επιτροπή. Είπαν πως θα έχουμε νέα προγράμματα και δεν θα επικεντρώνεται το ενδιαφέρον μας μόνο στα ίδια διατροφής έχουμε πολλούς συναδέλφους που εργάζονται στα, στα εθνικά ιδρύματα για την Αγγλία και λένε ότι θα πρέπει να διατεθούν περισσότεροι πόροι για εξοπλισμό σύγχρονο. Για πέστε μας, τα προγράμματα της Ένωσης θα καλύψουν τα τεχνικά προβλήματα. Ευχαριστώ. Να προσπαθήσω να απαντήσω έτσι λίγο συνεκτικά. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις καταρχήν και τις ανησυχίες που εκφράσατε. Είναι αλήθεια ότι ο προϋπολογισμός είναι μικρότερος ε, από ό,τι θα θέλαμε εμείς οι διαχειριστές των προγραμμάτων, αλλά πάντως αυτό αποφασίστηκε μέσα από πολιτικές διαδικασίες και έπρεπε να συμβιβαστούμε με τον προϋπολογισμό του εβδόμου προγράμματος πλαίσιο. Α, δεν ε, σας ικανοποίησαμε, αλλά πάντως πρόοδος έγινε. Και έγινε ένας έντονος διάλογος ε, με την νυν Μάρε για τις προτεραιότητες ε, και για τη μετάφραση των αποτελεσμάτων είτε στη διαχείριση των τρεχουσών πολιτικών ή για προετοιμασίες νέων πολιτικών. Είναι μια συνεχιζόμενη διαδικασία και όλα επιδέχονται βελτιώσεων. Αυτό το ξέρουμε. Υπάρχουν όμως ήδη καταγεγραμμένες πρόοδοι. Ίσως ε, δεν ε, τα γνωρίζετε λεπτομερώς όλα αυτά τα θετικά. Το νέο χρηματοδοτικό πακέτο σίγουρα στοχεύει σε αυτή την τρύπα που υπάρχει, όπως είπατε, που θα μεταφράσει τα ερευνητικά αποτελέσματα σε πρακτικές λύσεις. Καμιά φορά πρέπει απλώς να διασφαλίσουμε ότι η ερευνητική έρευνα θα χωνευτεί καλά και θα παρουσιαστεί σε κατανοητή μορφή για να συμπεριλάβει και να εντάξει στα ίδια τα προγράμματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ήδη έχουμε προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και αν δείτε και μετέπειτα προγράμματα στο πρόγραμμα πλαίσιο θα δείτε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις συμμετέχουν όλο και περισσότερο. Θα ήθελα εδώ να αναφέρω επίσης ότι μία από τις δραστηριότητες που ε, προωθούμε στο τωρινό πρόγραμμα πλαίσιο, όχι με χρήματα αλλά περισσότερο με θεσμική ενθάρρυνση, είναι η συγκρότηση των τεχνολογικών πλατφορμών. Υπάρχουν δύο τώρα. Η μία αφορά την υδατοκαλλιέργεια, η άλλη είναι μια καινούρια η οποία αφορά την αλληλεία, προϊόντα αλληλείας. Ε, λάβαμε υπόψη μας τον κλάδο και τα συμφέροντά του και έχουμε τώρα ένα feedback για τις προτεραιότητές τους. Είναι χρήσιμοι αυτοί οι μηχανισμοί και εις ό,τι αφορά την τροφοδότηση πληροφοριών για να μεταφράσουμε εμείς τις, προ... Ε, προτεραιότητες, αλλά και έχουμε μια διαμεσολάβηση, αν θέλετε, ούτως ώστε τα ερευνητικά αποτελέσματα να ξαναγυρίσουν στον κλάδο και να γίνουν γνωστά δεν μπορώ να σας δώσω νούμερα, γιατί ακόμα προφανώς δεν ξέρουμε ποιος θα είναι ο συνολικός προϋπολογισμός για αυτό το ερευνητικό χρηματοδοτικό πακέτο, το οποίο θα το παρουσιάσει η Επίτροπος στις 29 Ιουνίου, από ό,τι καταλάβαμε. Το συνολικό πακέτο σίγουρα πόρο απέχει από το να έχει ήδη αποφασιστεί και προφανώς θα περάσει χρόνος μέχρι ότου γίνει η κατανομή των κονδυλίων σε κάθε τομέα. Να πω όμως ότι είναι πιθανό ότι θα, αυτό το κοινό ε, επιστημονικό πρόγραμμα που χρηματοδοτήσαμε θα πρικοδοτηθεί αρκούντος και θα βρεθεί και εύκολος τρόπος για να συμμετέχει ο κλάδος, η βιομηχανία είτε από την αρχή, στη διάρκεια ή μετά. Θα υπάρχουν κάποιες δυνατότητες αναδιάρθρωσης. Ε, αυτές είναι οι υποδομές ερευνητικές, δεν είναι δηλαδή αλληλευτικών εργαλείων και υποδομής. Τα δύο, οι δύο τεχνολογικές πλατφόρμες θα παίξουν το ρόλο τους και αυτές και υπάρχει και ένα νέο στοιχείο το οποίο τώρα το σχεδιάζουμε και είναι ενδεχομένως μια πρωτοβουλία κοινή για τον προγραμματισμό που θα εξετάσει θέματα που αφορούν στους ωκεανούς. Αυτό είναι μια προσπάθεια συντονισμού από τα κράτη-μέλη, αλλά θα συμμετέχει προφανώς και η Κομισιόν, διότι και θα φροντίσει ώστε αυτή η συμπληρωματικότητα των δραστηριοτήτων να είναι δεδομένη και να διασφαλίσει και την ύπαρξη συνεργειών μεταξύ των διαφόρων μηχανισμών. Σαφώς όμως ε, δεν μπορούμε σε αυτή τη φάση να πούμε πολλά περισσότερα σχετικά με τα κονδύλια που θα διατεθούν είτε για όλο το χρηματοδοτικό πακέτο και σίγουρα όχι για τους επιμέρους τομείς που αυτό καλύπτει. Ε, ε άκουσα και μια ερώτηση για την υποστήριξη σύγχρονων εξοπλισμών. Συνήθως δεν γίνεται αυτό μέσα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος πλαίσιο, αλλά υπάρχουν περιφερειακά κονδύλια, διαρθρωτικά κονδύλια αν, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν αν επιτοπίως υπάρχει σχετική επιθυμία. Όταν γίνεται κοινή έρευνα, στηριζόμαστε στην υπόθεση ότι κάποιοι εξοπλισμοί που είναι βασικοί είναι διαθέσιμοι. Πρόσθετοι εξοπλισμοί μπορούν να συμπεριληφθούν αν το επιτρέψει ο προϋπολογισμός σε όλο το επιλέξιμο κόστος. Αλλά αυτά θα πρέπει να είναι εξοπλισμοί που αφορούν στην έρευνα, όχι γενική υποδομή. Για την απλούστευση, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι αυτό είναι μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζαμε επί πολλά έτη. Κάποια πρώτα βήματα έκανε η Επίτροπος και νωρίτερα μέσα στο χρόνο, στις 24 Ιανουαρίου συγκεκριμένα, ε, παρουσιάσαμε αρκετές απλοποιήσεις όσο μπορούσαμε χωρίς να γίνουν μεγάλες ε, νομικές αλλαγές, νομικές βάσεις που θα άλλαζαν που δεν ήταν δυνατόν να γίνει εκείνη τη φάση. Περαιτέρω αλλαγές ε, απαιτούν όμως μίζονες νομοθετικές αλλαγές που διέπουν τα σχετικά προγράμματα. Οπότε θα τις υποβάλουμε ως πρόταση αργότερα μέσα στο χρόνο και επίσης κάποιες μεγάλες αλλαγές, ίσως το ακούσατε και από άλλες επιτροπές, κάποιες μεγάλες αλλαγές που θα πλουστεύσουν τα πράγματα θα είναι αλλαγές στο δημοσιονομικό κανονισμό, διότι αυτό προκαλεί έναν αριθμό δυσκολιών, δηλαδή είναι υπερβολικά άκαμπτος ο δημοσιονομικός κανονισμός. Αν μπορέσουμε να τα αλλάξουμε αυτό αλλά σε υψηλό, σε ανώτερο επίπεδο, τότε θα έχουμε θετικές επιπτώσεις ε, στο επίπεδο της διεξαγωγής των ρυθμίσεων για τη χρηματοδότηση της έρευνας τα αποτελέσματα από το ερωτηματολόγιο, η συμβολή των οργανώσεων οργανισμών που αποκρίθηκαν, θα οδηγήσουν σε περαιτέρω απλουστευτικές ιδέες, ιδέες απλούστευσης, απλοποίησης και είπαμε ότι ένα σημαντικό πράγμα, ιδιαίτερα σημαντικό, αφορά τους τρεις τύπους των μέσων που προσπαθούμε να εντάξουμε σε αυτή την, υπό την αιγίδα του στρατηγικού πλαισίου για να έχουμε πιο τυποποιημένους κανόνες που δεν υφίστανται αυτή τη στιγμή ε, για να καλύπτουν τα χρηματοδοτικά πακέτα. Ε, θα έχουμε μάλλον περισσότερα ε, ε κατά ποσά από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα αλλά ελπίζω ότι γενικά θα διευκολυνθεί μέσα από ε, περαιτέρω προδιαγραφές ή χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη επακριβέστερα το κόστος. Αν μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε κατά αποκοπήν ποσά, αυτό θα απλουστεύσει πολύ τη διαδικασία. Η χρηματοδοτηση λαμβανοντα υποψη επακριβεστερα το κοστος αν μπορεσουμε να χρησιμοποιησουμε κατα λόγη για τη συνθετότητα σε αυτό το τομέα ανάγεται στο θέμα της λογοδοσίας. Ε, οι δημοσιονομικοί κανονισμοί πρέπει να το λάβουν υπόψη αυτό. ελπίζω να απάντησα. δεν απάντησε κυρία Πρόεδρε κάτι, πείτε μου. Σας ευχαριστούμε. Κύριε Βαλέσα, θέλετε να ολοκληρώσετε, θέλετε τώρα και πάλι τον λόγο. Να έχετε τον λόγο. No, dziękuję bardzo jeszcze raz panu przedstawicielowi komisji. Oczywiście to, co w tej chwili usłyszeliśmy, e, nie jest za e, Ευχαριστώ πολύ. Δεν μας ικανοποιεί η απάντηση του εκπροσώπου τη Κομισιόν βέβαια, αλλά ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά η αλληλεία και τα θέματα που μας ενδιαφέρουν δεν θα παραγνωριστούν όπως παραγνωρίστηκαν από το προηγούμενο πρόγραμμα πλαίσιο. Πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνει αυτό αυτή τη φορά και κάποια κονδύλια, κάποιες πιστώσεις να διατεθούν για την έρευνα στον τομέα το δικό μας. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε την Επιτροπή που θα μας μιλήσει και τον κύριο Βαλέσα και το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξή. Η συζήτηση του σχεδίου του κειμένου και υποβολή τροπολογιών 16 Ιουνίου, ψήφιση 12 Ιουλίου στην Επιτροπή μας και στην Ήτρε στις 30 Αυγούστου. Άρα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για να πάει στην Ήτρε. Σας ευχαριστούμε. Και έτσι Κλείσαμε το σημείο παριθμών 12. Πάμε στο 17ο τώρα. Παρουσίαση της μελέτης για τη γαρίδα στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτό ζητήθηκε από τους σοσιαλιστές. Να ευχηθούμε. Καλώς όρεσε Η κυρία Ντομινίκα Διάτ επιστημονική σύμβουλος της ε, AND. Και καλωσόρισε και ο κύριος Τόμας Νόιντέκερ του Ιδρύματος Γιώχαν Φον Τίνεν από τη Γερμανία. Όταν είστε έτοιμος, κύριε Βιάτ, έχετε το λόγο y cuando quiera usted tiene la palabra para explicar su informe. Merci, Madame la Présidente. Pour commencer, je vous... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Δεν μπόρεσε να έρθει και ζητήσει συγγνώμη μέσω εμού ο συνάδελφος γιατί έχει κλείσει το αεροδρόμιο του Αμβούργου. Επομένως, θα κάνω εγώ την παρουσίαση. Για να δούμε Γιατί έγινε αυτή η μελέτη. Ζητήθηκε για τέσσερι λόγου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρώτα-πρώτα, διαπιστώθηκε ότι η γκρίζα γαρίδα ως κλάδος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Υπάρχουν προβλήματα σε διάφορα κατημέλη. Επίσης υπάρχει ένα θέμα, μια στους προβληματισμός οικολογικός για το, για ποιες είναι οι επιπτώσεις της αλλίας επί του περιβάλλοντος. Τρίτον, έχουμε την μεταρρύθμιση της κοινής οργάνωσης αγοράς και της ε, κοινής πολιτικής, γιατί χτυπήθηκε ο κλάδος όσον αφορά την ε, καταγγελία της ε, Ολλανδικής Αρχής επί του ανταγωνισμού καταγγελίες κατά των βασικών συντελεστών του κλάδου. Επομένω, πρόκειται πάρα πολύ σημαντικό κλάδο σε, σε τρει χώρε, σε κάτω χώρε, Γερμανία και Δανία. Οπότε γι' αυτό και ζητήθηκε να διατυπώσουμε εμεί ένα ενημερωτικό έγγραφο, ενημερωτικέ προτάσει τα θέματα παραγωγή, τα θέματα θέση σε εμπορία, καθώ και τι εφαρμοστικέ λεπτομέρειε τη κοινή οργάνωση αγορά. Θα μόνο σε αυτή την παρουσίαση όσον αφορά ε, αυτέ τι τρει απόψει του θέματο και τι σχετικέ συστάσει. Η παραγωγή κρατά εδώ και μια τεσσαρκονταετία. Έχουμε νοδικές τάσεις, γιατί είχαμε 12 με 13 τόνους δεκαετία του 70, τώρα όμως που έχουμε ανέβει στους 35.000 τόνους και 40.000 για το 2010. Οι εκφορτώσεις γίνονται κυρίως σε τρία κράτη, Ε, Γερμανία 5% και κάτω χώρε και Δανία, Βέλγιο, Ενωμένο Βασίλειο και Γαλλία 5%. Η Δανία βασικά κινείται που είναι ο πιο μικρός τόλος στα χωρικά της ύδατα, η Γερμανία στις ε, δανέζικες γερμανικές αρχές ε, και βορείως των κατοχωρών και ο ο Ολλανδικός αλλιεύει παντού όπου υπάρχει γκρίζα γαρίδα. Η οικονομική και κοινωνική σημασία τώρα έχουμε 500 σκάφη και πάνω από χίλιους ναυτικούς οι οποίοι εμπλέκονται 500 είναι σχετικές συγκρίσεις ή άδειε που έχουν χορηγηθεί για την ελεία της ε, Γαρίδας Έχουμε δύο δημοκρατίε, δημοκρατίες, ε, κάτω Σαξονία, στο Χολστάιν και τη Γερμανία και τη Δανία. Έχουμε επίση 7 εκατομμύρια ευρώ μόνο για την Δανία στον αφορά εισόδημα. Αυτό είναι 2% του συνολικού εισοδήματο για το, το, τον αληθικό κλάδο γενικότερα στην Δανία και 68 είναι απασχολούμενοι και 3 τα σχετικά ε, λιμάνια και το λιμάνι που κυρίω χρησιμοποιείται είναι το Έσπιον. Στη Γερμανία βέβαια τα πράγματα είναι μεγαλύτερη τάξη μεγέθου διότι πάμε για 33 εκατομμύρια ευρώ ω ε, εισόδημα, 20% ε, του συνόλου των αλληλευτικών εισοδημάτων, 580 είναι οι επασχολούμενοι. Και στα δύο λάντρε που είπαμε, συνολικά έχουμε 580, 21 τα λιμάνια που χρησιμοποιούνται και έχουμε και 5 λιμάνια όπου ε, είναι πρωταγωνίστρια η Γαρίδα και αποτελεί και πόλο που τουριστικής έλξης στις κάτω χώρες. Επίσης, εκεί έχουμε το πιο ψηλό εισόδημα, 44 εκατομμύρια ευρώ, 14% του συνόλου των ε, εισοδημάτων από την θαλασσία αλληλεία όπως ε, είχα τη Γερμανία και εδώ έχουν περίπου 500 και 7 είναι τα λιμάνια τα οποία χρησιμοποιούνται τα περισσότερα ε, στο, στο βόρειο κομμάτι της χώρας ε, τώρα όσον αφορά την δομή, τη διάρθρωση του στόλου της κάθε χώρας. Ο πιο μικρός είναι ο Δανέζικος, αλλά είναι και ο πιο σύγχρονος. Είναι η πιο αποτελεσματική πολιτική αλληλεία στην Δανία, στην ε, Γερμανία. Έχουμε πάρα πολλά μικρά αλλά και παλαιά σκάφη. Υπάρχει εποχιακός χαρακτήρας όσον αφορά τον τρόπο αλληλείας. Στις κατοχωρές έχουν ε, τα πιο σχεδόν μοτέρ, τα σκάφη και εκφορτώσεις είναι πιο μεγάλες και άλλωστε όλη τη χρονιά και συνέχεια αλλιεύουν αυτά τα σκάφη. Τώρα όσον αφορά την αποδοτικότητα για αυτή την αλία, να σας τα πω εδώ εντάχει. Έχουμε εδώ τρεις γραφικέ παραστάσει ε, και διαπιστώνουμε ότι στην Δανία η αποδοτικότητα εξασφαλίζεται συνεχώ όλα αυτά τα χρόνια τα οποία εδώ εξετάζουμε, το 2002 δηλαδή μέχρι το 2008. Και διαπιστώνεται ότι ε, αυτή η αποδοτικότητα ε, είναι ευθέω ανάλογη με την τιμη πώληση πώλησης. 10-11 έχουμε πτώσει και επομένω είναι επιζήμια η κατάσταση για το, το στόρο στη Γερμανία, η αποδοτικό της ε, ήταν μέχρι το 2007 ασήμαντη, όμως πήγαν κάτι από το 2008 γιατί ανέβηκαν οι τιμές αλλά είχαμε κατακρίμηση της τιμής 9, 10 και αρχές του 11. Βλέπετε και εδώ επομένω ότι ακολουθήθηκε η ίδια διαδρομή και για τις κάτω χώρες όσον αφορά τις ε, συνθήκες ε, διαπιστώθηκε ότι δεν είναι σίγουρη αποδοτικότητα ε, και στις τρεις αυτές χώρες έχουν κάνει απεργία οι ψαράδες δύο απόπειρε γίνονται τόσο ώστε να εξασφαλιστεί η αποδοτικότητα. Πρώτα-πρώτα ε, στο Βάγγενιγκεν έγινε μια πρωτοβουλία για να εξασφαλιστεί ε, μια αποδοτικότητα σταθερή. Είπαμε ότι πάμε σε πρώτη τιμή πώληση 2,25 μεταξύ 25 και 3 και 50 ε, κινείται η τιμή ανάλογα με την εποχή, ανάλογα με τη ζώνη, με τη χώρα. Οπότε μόνο εάν η τιμή είναι πάνω από 3,5 ευρώ το κιλό, μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μακρόπνη, μακροπρόθεσμη αποδοτικότητα. Βλέπετε μετά, σε αυτό το στριμωγμένα της διάκριτα λέει ο, ο πίνακας, προσπαθεί να δει ακριβώς ε, το ακαθάριστο κέρδος πώς διαμορφώνεται βάση για αυτόν τον πίνακα είναι η κατανάλωση του ντίζελ 1,67 ε, ανά ε, ψαρά 54.000 είναι το κόστος ανά σκάφος και βλέπουμε επίσης ότι μόνο από 58 και πάνω πάνω πει ότι θα υπάρξει μακρόπνοη αποδοτικότητες. Μεταξύ Νοέμβριο και Φεβρουάριο εκπονήθηκε αυτή η στατιστική. 55 σαντίμ ήταν η τιμή του ντίζελ τότε. 0,70 είναι το κόστος. Και 2,58, 2,60 ήταν η τελική τιμή. Στην δεξιά βλέπετε τι θα γίνει εάν έχουμε μείωση από 500 σε 375 σκάφη, μείωση του στόλου. Και βλέπουμε το νεκρό σημείο από το οποίο αρχίζει η αποδικότητα είναι στα 42-43 σαντίν για το στόλο των 500. Τώρα τι γίνεται με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, εκείνες οι οποίες ε, ασχολούνται εξειδικευμένα με τα θέματα του περιβάλλοντος, λένε ότι το παραλίευμα και τα, τα, οι απορρίψεις δημιουργούν πρόβλημα στη θάλασσα. Απορρίψεις. Και τα παραλίευματα θα παρεμπίπτονται. Ε, επίσης, είπαμε όμως εδώ δεν έχουμε κάποιο είδου δείγματα υπεραλήψης που είναι καλά η αληθική πόρη. Εδώ το 14 εξαρτάται από την θερμοκρασία. Ο Μερλούκιος ε, έχει αρνητική επίδραση γιατί κυνηγάει τη γαρίδα. Και τέλος τα παρασυρώμενα δίχτυα οι τράτε έχουν αρνητική συνέπεια. Συγγνώμη, δεν έχουν συνέπεια όσον αφορά το βυθό. Τελευταία σημαντική μελέτη όσον αφορά τις απορρίψεις έγινε από τον Ναπόντα συνάδελφο το 2006 στη βάση έκθεσης του 2005. είχαμε 38 χιλιάδες τόνους και πήγαμε στους 100 ε, και πετάχθηκαν πίσω στα άλλα 123.000 τόσες ε, γαρίδες πίσω στα άλλα και επομένως ε, πήγαμε στο 70% όσον αφορά το ποσοστό επιβίωσης. Μετά είχαμε μαγείρα με τις γαρίδες, βράση με γαρίδες πάνω στο σκάφος 58.000 τόνων και κατόπιν είχαμε δεύτερη διαλογή και απόρριψη νεκρές γαρίδες αυτές και κατόπιν μετά την αποβίβαση είχαμε εκφόρτωση 49.000 τόνων και κατόπιν είχαμε τρίτη διαλογή από τους χονδρεμπόρους και τους μεταποιητάς στην ξηρά. Και έτσι ε, βγαίνουν τις και φτάνουμε σε μια παραγωγή και θέση εμπορία 38.000 τόνων που είναι 21% του αλλιεύματος. Το σύνολο επομένως είναι 60% του αλλιεύματος αλλά 68% είναι 78% είναι η απόρρευση και 60% είναι το ποσοστό επιβίωσης και για μέσα έχουμε 18% που έχουν πεταχτεί λόγω θανάτου. Και επίσης βλέπουμε εδώ πέρα ότι βλέπετε αυτές οι τράτες τι επιπτώσεις έχουν ε, υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση που επισημαίνει ότι έχουμε εδώ δύο είδη τέτοιων ε, σκαφών άλλο για ψάρια και άλλο για γαρίδες και πρέπει να μια σύγχυση για τα επίπεδα ψάρια ε, είναι πιο βαριά η τράτα ενώ για τις γαρίδες είναι πολύ ελαφρύτερη από ό,τι για τα πλατήψαρα. Εκεί υπάρχουν κάτι, κάτι πράγματα σαν ροδάκια, ούτω ώστε να μπορεί να ρολάρει να σύρεται έτσι, πάνω στα ροδάκια, στο, στο βυθό αυτή, αυτό το, το δίχτυ, αυτό το εργαλείο ελίας. Και μπορεί να δείτε εδώ μια φωτογραφία για το πώς λειτουργεί αυτό το δίχτυ με αυτού του είδους τα ροδάκια για να μπορεί να προχωράει πάνω στο βυθό. Αυτά όσον αφορά τώρα το είναι, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, το βασικό πρόβλημα είναι ε, το, το, και τα, οι απορρίψεις. Δύσκολο να προχωρήσουμε με δίχτυα που έχουν τετράγωνα μάτια σε σχέση με τους ρόμβους, τους παραδοσιακούς, γιατί έτσι μειώνεται το παραλίευμα όσον αφορά τα στρογγυλά ψάρια και τη μικρή γλώσσα. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια μείωση δραστηριότητα από Ιούνιο μέχρι Αύγουστο. Γιατί τότε έχουμε το, τα μεγαλύτερα παραλίευματα. Και έχουμε εδώ κάποιο είδου έχουμε τέτοια δίχτυα εμφανίας κατά την, μεγαλύτερη περίοδο. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ε, εξαιρέσεις, τις οποίες θα πρέπει να εξαλείψουμε. Και θα πρέπει να αποφύγουμε να ψαρεύουμε στα ρίχα. Γιατί εκεί προκύπτει το μεγαλύτερο παραλίευμα. Όσον αφορά τώρα την διαχείριση του αλλιεύματος ή των πόρων, Υπάρχουν κάποια προγράμματα στα κράτη-μέλη. Αφορούν ώρες και διάρκεια αλίας, αφορούν τη, τη μείωση του αλλιεύματος, αφορούν ε, τα στοιχεία της δυνατότητας του σκάφους, καθώς και το παραλίευμα. Τώρα, οι αγορές. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι 34.700 τόνοι το 2010 όσον αφορά την εκφόρτωση. Βλέπετε εδώ μια παράσταση της αγοράς που δεν αντιστοιχεί με την παραγωγή. Γιατί το Βέλγιο καταναλώνει ως αγορά πάνω από τα μισά της συνολικής παραγωγής και δεύτερη έρχεται η Ολλανδία και η Γερμανία που επίσης έχουν σημαντικό κόμμα κατόπιν η Γαλλία με 7% είναι πολύ σημαντικό σημαντικός τη ε, ολόκληρων, μη αποφλειωμένων γαρίδων η Γαλλία. Οι τη αγορές πάνε στην αποφλειωμένη και οι υπόλοιπε χώρε στην Ευρώπη είναι το 3% τώρα. Το βασικό χαρακτηριστικό τη αγορά είναι η συγκέντρωση. Είναι μόνο δύο οι εταιρείε ε, Ολλανδικέ που κατέχουν το 80% του μερίδιο τη αγορά, High Plug και Class Pool και επίση μένει το 20% όσον αφορά ε, διάφορους χονδρεμπόρους και με, μεταποιητάς οι οποίοι και αυτοί είναι όμως όσο το πλήστον Ολλανδοί. Δυο λόγια τώρα για την καθεμία από αυτές τις αγορές των τριών χωρών στη Δανία. Δεν έχουμε σημαντική αγορά στη Δανία, δεν ε, ασχολούνται άμεσα με το τι γίνεται στα ε, λιμάνια. Οι Δανείοι ούτε κάνουν την μεταπίση γιατί την έχουν λάβει οι Ολλανδικές εταιρείε και επίσης ασχολούνται με τι Σκανδιναβικέ, με την Ιρλανδία. Ε, και επίση κάνουν και τι θέσει έχει σταματήσει η θέση εμπορία της κυρία Γαρίδα. και επομένω οι περισσότεροι που ασχολούνται είναι οι Ολλανδοί στην Δανία και κάνουν τη μεταποίηση αφού μεταφέρουν στη χώρα του τη γαρίδα τη Δανέζικη. Τώρα η Γερμανία είναι η πιο μεγάλη αγορά, ε, είναι τη τάξη των 5.600 τόνων, περίπου 20 είναι κάποιε μικρέ ε, τέτοιε εξεδημένες επιχειρήσει, οι οποίε εξειδικεύονται όσον αφορά το χονδρεμπόριο αλλά και την μεταποίηση και θέτουν σε εμπορία στη χώρα του το προϊόν και υπάρχουν οι δύο βασικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη Γερμανία είναι η Highplug και η Pool που έχουν θηγατρικές ε, ή στην Γερμανία. Η Ολλανδική αγορά τώρα είναι κάτι σαν τη Γερμανία ως αυτό το μέγεθος. Ε, μιλάμε για 5.700 τόνους. Έχουμε δύο, βασικές, λοιπόν δύο βασικές εταιρείες, η Hybrid και η Class Pool, που αγοράζουν περίπου και οι δύο 30.000 τόνους γκρίζας γαρίδας. Η δε γκρίζα γαρίδα στον τζίρο αυτών των εταιριών αντιστοιχεί στο 30% για κάθε εταιρεία. Και έχουμε επίσης την ε, Haiko και την Telson και αυτές ε, Ολλανδικές που εμπλέκονται. Η Haiblock είναι πάντως ο πρωταθλητής της αγοράς, ο μεγαλύτερος προμηθευτής. Στο Zoutkamp έχει το μεγαλύτερο εργοστάσιο μεταποίησης. Μιλούμε για 250 εργαζομένους. Έχει επίσης και θηγατρική που κάνει την μεταφορά. Φορτηγάκια τα οποία πάνε και έρχονται προς και από το Μαρόκο για αυτή την αποφλίωση που, την οποία έλεγαν προηγουμένως αλλά γίνεται έτσι και η διανομή του τελικού προϊόντος στις διάφορες αγορές. Επίσης, στη Γερμανία έχουμε την Bizumer Fischerei. 70 από τους 80 ε, τους απέλησε. Πήρε σε αστυνοτά η Goldfish της κατοχώρας επίσης. Και αυτοί, επομένως, ε, απευθύνονται στο εργοστάσιο του και επίσης και αυτοί αναφέρουν στους Μαροκινούς την αποφλίωση. 70% είπαμε. 70% ε, είναι οι πωλήσει στο, στο Βέλγιο. Η ΔΕ. Ε, Χαϊπλούχ. και οι Μπούζουμερ στη Γερμανία. Κάνουν την διαλογή αλλά και την ε, ε, συσκευασία των προϊόντων που μετά πάνε στις κάτω χώρες. Και η, και η Κλασπούλ κάνει ε, με τους Μαροκινούς την αποφλίωση επίσης. Ολλανδοί και Γερμανοί έχουν προσπαθήσει τοπικά σε κάτω χώρε και η Γερμανία να γίνεται η αποφλίωση και να γίνεται και με τρόπο μηχανικό. Όμως η απόπειρα του απέτυχε πέρσι δε. Προσπάθησε μια εταιρεία σε μεγάλη κλίμακα να εφαρμόσει αυτό το μηχανικό τρόπο αποφλίωσης. Πρόβλημα ήταν το ότι μηχανικά δεν είναι η αποφλήση το ίδιο ποιοτική όσο με τα χέρια. 28 σε σχέση με το 2% επίσης είναι το αποτέλεσμα. Και επίσης κοστίζει πάρα πολύ. Επομένως, έχουμε την Χάιπλουχ, η οποία βέβαια συνέχισε να συναλλάσσεται με πάρα πολύ εξειδικευμένη βιομηχανία στις ε, χώρες και επομένως σαν μέσο όρο είπαμε ότι κρατάει 15 μέρες αυτή η διαδικασία της αποφλίωσης και όλοι τελικά δουλεύουν με το Μαρόκο. Στο Τετουάν είναι 1400 εργαζόμενοι στη Χάιμπλουχ και είναι και άλλοι τέσσερις υπεργολάβοι ούτως υπήρχε στο Μαρόκο. Η Χάικο και η Τέλσον επίσης έχουν κάποιους που δουλεύουν στο Μαρόκο για αυτούς. Το δε κόστος που τους αποκλείσουν είναι 5,20 ευρώ ανά κιλό. Τούτο για να δούμε τώρα ποιο είναι το περιθωριό κέρδος, ποιες είναι οι τιμές. Έχετε εδώ τις ε, τιμές που αφορούν τον Ιανουάριο του 2011. Έχουμε μια μέσα τιμή ανά κιλό ε, εκφόρτωσης των ύψους 2 ευρώ, 33 εκατοστά ε, μήκος και φτάνει στα 2,33 ευρώ για τους χονδρεμπόρους επί τρία, διότι απαιτούνται τρία κιλά ε, γαρίδες που εκφορτώνονται για να παραθεί ένα κιλό φλοιωμένο. Ε, σας είπα για το κόστος της αποφλίωσης και τελικά ε, το η αποφλοιωμένη γαρίδα φτάνει τα 12,19 ευρώ. Τιμή πώλησης ε, των μεταποιητών ε, ανερχόταν το Ιανουάριο του 2011 μεταξύ 17 και 25 ευρώ, ενώ η τιμή αγοράς ήταν μεταξύ 21,10 και 39,90 ευρώ ανάλογα με το μέγεθος και τον τρόπο διανομής. Στη δεξιά στήλη του πίνακα βλέπετε τους υπολογισμούς που έχουν γίνει επί τη βάση μιας τιμής 3,5 ε, ε, ευρώ ανά κιλό, δηλαδή η τιμή ε, όταν φτάνει στον μεταποιητή και μετά αφού γίνει η επεξεργασία το κιλό φτάνει στα 16,69 ευρώ. Και διατηρείται η τιμή κοντά στο κόστος. Τώρα, η εικόνα, που, η εικόνα στον καταναλωτή της ε, γαρίδας είναι καλή η εικόνα. Ε, οι περισσότεροι προτιμούν δηλαδή την ε, γκρι γαρίδα σε σχέση με την ροζ γαρίδα. Μπορούμε να πούμε επίσης ότι οι καταναλωτές γενικώ δεν γνωρίζουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα της γαρίδας, δηλαδή οι περισσότεροι αγνοούν την μακρά ε, πορεία που διανύει η γαρίδα και φτάνει στο Μαρόκο για να ξαναγυρίσει πίσω στην Γερμανία και γίνεται και μάλιστα και μία ανάμιξη ε, νοπών και κατεψυγμένων δεν γνωρίζουν οι καταναλωτές επίσης το πώς γίνεται η συντήρηση και το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αλίευσης και της ε, τελικής πώληση στην αγορά. Τώρα, ε, οι θέσεις των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Τώρα στα θετικά στοιχεία είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τα ίδια αυτά. Θα μπορούσα να πω δύο λόγια σχετικά με την διαδικασία η οποία δρομολογήθηκε από, τις Ολλανδικές, από την Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού, διότι πρόκειται για μια διαδικασία και η, η τελική διευθέτηση είναι πολύ πρόσφατη, πριν από τρεις μήνες. Ε, και ακριβώς αυτό επηρεάζει και τους ε, εμπλεκόμενους στον κλάδο και την αγορά. Έτσι λοιπόν ε, έγινε μια δικαστική διαδικασία εναντίον των παραγωγών, των οργανώσεων παραγωγών και των χονδρεμπόρων με την καταγγελία ότι παραβίασαν τους κανόνες ανταγωνισμού τους κατηγορούσαν ότι καθόριζαν ελάχιστη τιμή αλλά επίσης και περιορισμούς ε, πέραν της ε, ε, τριμερούς συμφωνίας στο διάστημα 1η Ιανουαρίου 1998 έως 30 Ιανουαρίου 2010 και βεβαίως η συμφωνία αυτή είχε ως στόχο να παρεμποδίσει την εισαγωγή στην αγορά νέων εμπόρων. Έτσι λοιπόν ελήφθη μία απόφαση για οκτώ ε, φορείς και οκτώ χονδρεμπόρους και το εφετείο τον Δεκέμβριο του 2004 ε, διέκοψε τις, ε, τα πρόστιμα για τους μικρούς παραγωγούς και μείωσε τα πρόστιμα για τους υπολείπους σε 6,2 εκατομμύρια. Το Δεκέμβριο του 2006 μειώθηκαν ακόμα περισσότερο τα πρόστιμα σε 5,4 εκατομμύρια και η ανώτατη αρχή, η οποία ήταν υπεύθυνη για την τελική διευθέτηση ε, στο πλαίσιο του ανταγωνισμού η ΣΕΜΠΕ έλαβε την οριστική απόφαση στις 22 Μαρτίου του 2011 και τελικά τα πρόστιμα που πρέπει να καταβληθούν ανέρχονται σε 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν μειώθηκαν όπως βλέπετε επανειλημμένως και αυτό επειδή υπήρξε αυτή η διαφορά μεταξύ των παραγωγών και των χονδρεμπόρων. και ακριβώς επειδή η ΕΝΕΜΑ έλαβε υπόψη το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις των τριών χωρών ήταν υπέρ των ε, δεσμεύσεων που είχαν αναλάβει οι εταιρείε έναντι της ΠΣΠ και της ΟΣΕΜ ούτως ώστε να εφαρμοστεί η κοινοτική νομοθεσία. Ότι δηλαδή δεν πρέπει να καθορίζονται ελάχιστε τιμέ. Και ε, σε αυτό στο οποίο είχαν καταλήξει τριμερείς ε, διαπραγματεύσεις. Έτσι λοιπόν η ΕΝΕΜΑ αποφάσισε να παρακολουθήσει με μόνιμο τρόπο τον κλάδο της Γαρίδας στην Ολλανδία και το εφεξής η οι έμποροι και όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί ως προς τη διακίνηση της γαρίδας. Και τώρα θα έρθω για θα σας μιλήσω τώρα για την κοινή οργάνωση της ε, αγοράς, ε, λαμβάνοντας υπόψη τις ε, θέσεις των παραγωγών οργανώσεων. Υπάρχουν 27 ε, σκάφη που είναι οργανωμένες στην ε, Δανία. Στην Γερμανία η οργάνωση είναι ε, λιγότερο εύρωστη, 80%. Υπήρξαν τεράστιες αλλαγές, μειώσεις, κλείσιμο. Η τελευταία εξέλιξη ήταν το Δεκέμβριο του 2010. Έγιναν δύο συγχρονεύσεις, συγχωνεύσεις και έχουμε δύο βασικούς φορείς παραγωγής που συγκεντρώνουν το 74% των σκαφών και 81% της παραγωγής. Στην ε, Ολλανδία τώρα το ποσοστό οργάνωσης 90% υπάρχουν 7 φορείς ο βασικός είναι η Netherlands Fisher Bond και υπάρχουν και έξι άλλες εταιρείε, η κυριότερη εκ των οποίων είναι η Visnet. Τώρα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε ένα ποσοστό οργάνωσης αρκετά υψηλό, 88%. Εδώ πρέπει να προσθέσουμε ότι μια διεθνική οργάνωση παραγωγών συγκροτήθηκε το 2005 μετά από πρωτοβουλία της NMA της Ολλανδίας, ούτως ώστε να υπάρξει ρύθμιση της αλίας της Γαρίδας. Την 1η Ιανουαρίου 2011 αυτή η διεθνική οργάνωση εκπροσωπεί το ίμιση του στόλου. Η δράση των φορέων παραγωγών της Γαρίδας είναι αρκετά περιορισμένη επειδή υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ των διαφόρων ε, παραγωγικών οργανώσεων στην Ολλανδία και την Γερμανία και ε, εξαιτίας των ε, βασικών απαιτήσεων που βάζει η ΕΝΕΜΑ. Υπάρχει μια συζήτηση γενικότερα γύρω από το επάγγελμα στην Ολλανδία σχετικά με τις ποσοστώσεις. Το σύστημα ποσοστώσεων, δηλαδή υπάρχουν αλληλείς οι οποίοι θέλουν να υπάρξει σταθεροποίηση και των εκφορτώσεων και των αγορών, ούτω ώστε να υπάρξει μια ισορροπία στο περιβάλλον και τα αποθέματα και με αυτόν τον τρόπο δια διασφαλιστεί και μια σταθερότητα στην εμπορία και να υπάρξει και μια πιο σταθερή παρακολούθηση επιστημονική της ε, γαρίδας. Αυτοί που υποστηρίζουν τις ποσοστώσεις, την εισαγωγή ποσοστώσεων, λένε ότι αυτό θα διευκολύνει και την διαδικασία πιστοποίησης που είναι ευθύνη των ε, οργανώσεων παραγωγών. Αλλά υπάρχουν και διαφωνούντες μεταξύ των αλλιέων, αλλά και από πλευράς κεντρικής διοίκησης των ε, ε, χονδρεμπόρων και μεταποιητών που θεωρούν ότι πρόκειται για έναν περιορισμό της ελευθερίας που ισχύει στην αγορά και ότι αυτό καθιστά πιο δύσκολη την εισαγωγή νέων εισερχομένων. Και επίσης ε, όλοι αυτοί οι έλεγχοι είναι δαπανηροί και αν αυτές οι ποσοστώσεις εφαρμόζονταν θα υπήρχε ε, ο κίνδυνος συγκέντρωσης των εκφορτώσεων σε συγκεκριμένα σημεία και αυτό θα ήταν κάτι που θα έπλητε την Γερμανία. 18 Απριλίου 2011 η ΕΝΑΜΑ απέρριψε κάποιες προτάσεις που έκαναν οργανώσεις παραγωγών. Απέρριψε λοιπόν τις προτάσεις για τον περιορισμό αλίευσης με τα εξής επιχειρήματα. Πρώτον ότι δεν χρειάζεται να υπάρχουν τέτοιοι περιορισμοί δεύτερον ότι ο πληθυσμός της Γαρίδας δεν, είναι, δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο και επίσης ότι κάτι τέτοιο δεν επιτρέπεται από την Ολλανδική Αρχή Ανταγωνισμού. Ένα μέσο είναι η απόσυρση. Αυτό το εργαλείο, αυτό το μέσο, χρησιμοποιείται ελάχιστα ως προς τη Γαρίδα. Το 2009, παραδείγματο χάρη, που ήταν ένα σημαντικό έτος, ε, η απόσυρση εκπροσωπούσε το 0,66 των συνολικών εκφορτώσεων. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της ενιαίας οργάνωσης αγοράς, έγινε μια προσπάθεια ε, οργάνωσης. Οι Δανείοι θεωρούσαν ότι δεν χρειαζόταν μια τέτοια ε, διεπαγγελματική οργάνωση, διότι εκεί έπρεπε να συγκεντρωθούν οι αλληλείς, οι ε, απασχολούμενοι με τις υδατοκαλλιέργειες, οι μεταποιητές κλπ. Και να υπάρξει μια ενιαία ομπρέλα. Ε, θεώρησαν ότι μια συμβουλευτική επιτροπή είναι επαρκής. Στο πλαίσιο αυτής της μελέτης ε, τέθη το ερώτημα από την Επιτροπή Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζοντα ότι υπάρχουν ποσοστά ως προς τους δασμούς και αυτό αφορά τα 20, τους 20.000 τόνους, Ε, και το ερώτημα ήταν αν αυτό θα επηρεάσει την αγορά της ε, γκρίζας γαρίδας. Οι εμπλεκόμενοι συμφωνούν ότι δεν υπάρχει επίπτωση διότι η γκρι γαλίδα είναι απολύτω ανεξάρτητη. Τώρα, η πιστοποίηση MSC ε, που ισχύει στις τρεις χώρες μέλη. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σχέδια διαχείρισης που δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί και υπάρχουν κάποια κοινά σημεία, δηλαδή προσπάθειες βελτίωσης των τεχνικών αλίας, σχέδια μείωσης της αλληλευτικής προσπάθειας για να μειωθούν οι απορρίψεις και τα παρεμπίπτοντα ή παρελκόμενα αλλιεύματα. Από την άλλη, Υπάρχουν διαφορές ως προς την συνολική αλλιευτική προσπάθεια, δηλαδή το συνολικό αριθμό ορών ε, στην θάλασσα ανά και ως προς το αποδεκτό ε, μερίδιο μικρών γαρίδων στις εκφορτώσεις. Ε, δηλαδή στην ίδια ζώνη αλίας θα μπορούν να υπάρχουν τρία σκάφη με διαφορετικά βάρη. Τώρα, η πιστοποίηση αμεσέ δεν έχει οριστικοποιηθεί και πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από το 2012. Τώρα, τα βασικά συμπεράσματα στα οποία μπορεί να καταλήξει κανείς. Δηλαδή, τα αποθέματα είναι σε καλή κατάσταση, δεν υπάρχουν σημάδια υπεραλίευσης, η αλίευση ε, γκρίζας είναι πολύ σημαντική για τους στόλους της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Τα, οι τράτες 12 ε, 24 μέτρα της Γερμανίας και της Ολλανδίας εξαρτώνται απολύτως από την αλίευση της Γκριγαρίδας η τιμή για να είναι αποδοτική δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη από 2,75 ευρώ ανά κιλό. Η κατάσταση έχει ε, χειροτερεύσει πολύ αισθητά τους τελευταίους μήνες με διάφορες απεργίες που έχουν γίνει από τους αλλοί στην ε, Βορεια Θάλασσα. Υπάρχει μια υπέρ χωρητικότητα του στόλου υπέρ ε, διάθεση ε, ποσοτήτων στην αγορά. Η εφαρμογή της ενιαίας οργάνωσης αγοράς ε, έχει μικρή επίπτωση στην αγορά της γκριγαρίδας. Υπάρχουν εσωτερικές διαφωνίες μεταξύ Γερμανών και Ολλανδών ε, αλλιέων ως προς τις ε, βασικές αρχές της ΕΝΕΜΑ υπάρχει ισχυρή συγκέντρωση, συγκέντρωση σε συγκεκριμένα σημεία των φορέων επεξεργασίας και μεταποίησης και βεβαίως ε, οι λιανικές τιμές είναι εξαιρετικά κερδοφόρες για τους φορείς επεξεργασίας και λιανικής πώληση. Έτσι λοιπόν, οι συστάσεις είναι καταρχήν να γίνουν προσπάθειες ώστε να μειωθούν οι απορρίψεις και τα παρεμπίπτοντα αλλιεύματα. Να ενισχυθεί η έρευνα για ε, την ανάπτυξη νέων τρατών ε, που θα έχουν μειωμένη κατανάλωση καυσίμου αλλά και ε, μειωμένες απολύψεις ε, να εξεταστεί η μείωση του στόλου σε συνδυασμό με τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις, να διευρυνθεί το ζήτημα, η όλη συζήτηση σχετικά με τα συνολικά επιτρεπόμενα αλλιεύματα, τα TAC, ε, να υπάρξει σημαντική βελτίωση ως προς την ποιότητα με την ε, και εφαρμογή ε, κωδίκων δεοντολογίας από πλευράς αλλιέων ε, και επίσης να επιταχυνθεί η διαδικασία πιστοποίησης MSC. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον φορέα που εκπώνησε την έρευνα αυτή, η οποία ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένη, ακριβής και λεπτομερής. Και Τώρα θα ήθελα να ανοίξουμε την συζήτηση και όσοι επιθυμούν παρακαλώ να λάβουν το λόγο επί του θέματος αυτού. Παρακαλώ κυρία Λεβίνα να έχει το λόγο. Είναι η πρώτη που ζήτησε το λόγο. Κυρία Λεβίν. Ε, thank you very much. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόβιν γιατί είναι πάρα πολύ συναρπαστική η παρουσίαση που ακούσαμε για, για την κρίση Ζαχαρίδα, για το 80%, το παραλίευμα, για το τι γίνεται με το ξεφλούδισμα και για το πώς έχουν τα πράγματα στην αγορά. Τι γίνεται μέχρι να φτάσει στα χέρια, στα τραπέζια του καταναλωτή, γεμάτη με συντηρητικά. Δεν ξέρω πού να ξεκινήσω. Ήταν πάντως πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά, γιατί εγώ δεν γνώριζα καθόλου ότι στην Ευρώπη τη σήμερα ημέρα ανεχόμαστε τον, έχουμε 182.000 τόνους που αλλιεύονται ούτως ώστε να, να, να πουλήσουμε 38 και να πετάμε το 18 το, το 80 Φυσικά και υπάρχουν τα μέσα να αποφεύγουμε το παραλίευμα. Έχουμε αυτά τα τετράγωνα δίχτυα, τα τετράγωνα ματάκια τέλος πάντων. Άρα μπορούμε να αποφύγουμε αυτά τα ονομαζόμενα παραλίευματα. Είναι ντροπή. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε μόνο δύο εταιρείε οι οποίε θησαυρίζουν για από αυτό το 80% κομμάτι τη αγορά που έχουμε. Αυτέ που κατονομάστηκαν. Αυτές λοιπόν πρέπει να αναλάβουν ευθύνη. Αυτές φέρουν την ευθύνη, διότι βγάζουν τεράστια κέρδη από τους κοινούς πόρους της φύσης και για το μέλλον της αλίας των θαλασσίων ειδών, για το μέλλον του, περιβάλλον, το μέλλον του περιβάλλοντος, ε, πρέπει να περιοριστεί αυτή η ε, πέσχυντη συμπεριφορά. Έχω και κάποιες ερωτήσεις. Είπατε ότι το ποσοστό επιβίωσης των απορρίψεων φτάνει και στο 60%. Και αναρωτιέμαι, ποια είναι αυτά τα παραλιεύματα, τα παρεμπίπτοντα, τι είναι, ποια είναι τα κυρίαρχα είδη εκεί και πώς καταλήγετε στο 60% γιατί συνήθως μιλάτε όχι, 16%. Γιατί μιλάτε για 5% ή 1% συνήθως επιβιώνουν. Οπότε πώς επιβιώνουν αυτοί, αυτά τα είδη σε τόσο υψηλό ποσοστό. Μάλλον 16 πρέπει να εννοεί. Επίσης, ε, κάτι άλλο που μου κίνησε την περιέργεια. Στην παρουσίασή σας λέτε πώς τα ποσά προσθέτουν το κόστος της, γα... Ε, ε, γαρίδας για τον καταναλωτή. Και η αφαίρεση του κελίφους της γαρίδας, αν θυμάμαι καλά είπατε ότι είναι κάπου 3 ευρώ το κιλό, κάτι τέτοιο, είπατε. Αλλά η μεταποίηση η μεταποιητική βιομηχανία παίρνει δηλαδή καθαρισμένη τη γαρίδα και παρόλα αυτά προσθέτει 5 με 10 ευρώ και εκείνη το κιλό τη γαρίδα. Οπότε να ρωτιέμαι, αυτοί τι κόστος έχουν ως μεταποιητική βιομηχανία για να φορτώσουν απάνω στη γαρίδα αφού η γαρίδα έχει ήδη ε, καθαριστεί από το κέλυφος όταν αυτοί το παίρνουν, όταν αυτοί παίρνουν το προϊόν. Επίσης, είδα τις αξιολογήσεις της γαρίδας που, δε, που είναι ε, καλές, αλλά εξαρτάται και από άλλα είδη που την κυνηγούν. Και αναφερθήκε, ας πούμε, ο γάδος. Υπάρχουν τόσες πολλές τέτοιες γαρίδες, γιατί είναι λίγα τα είδη που κυνηγούν τη γαρίδα αυτή. Επίσης, ο Ολλανδικός νόμος περί ανταγωνισμού που δεν επιτρέπει την επιβολή φόρου, ε, που δεν, που δεν ε, επιτρέπει τάκ, ε, συνολικά ανώτατα επιτρεπόμενα αλλιεύματα. Άμα επιβάλλονται από την πολιτική αλλίευση, τι δουλειά έχει η πολιτική ανταγωνισμού. Εσείς μιλήσατε για εθελοντική, φαντάζομαι ότι αναφερόσαστε όχι στα επίσημα τάξ της Ένωσης, αλλά σε προαιρετικά ανώτατα επιτρεπτά αλλιεύματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, λέει κυρία Ρότς. Λυπάμαι που δεν μπορεί να είναι εδώ ο κύριος Νόιτακερ σήμερα. Έπεσε θύμα της ε, ηφαιστειακής τέφρας ε, που δεν, του, ε, δεν επέτρεψε Η μελέτη του κυρίου Νόιντεγκερ από το 2005 τώρα πάντως βελτιώνεται, επικαιροποιείται και θα έχουμε καινούρια δεδομένα εις ό,τι αφορά την αλληλεία. Εγώ είμαι από το Σλέσφιχ Χολστάιν και γνωρίζω και προσωπικά πολλούς που έχουν τράτες υπάρχουν, οι καθαρές τράτες που δεν έχουν ε, σχέση με... Ε, ε, ξέρω πολλούς ε, που αλλιεύουν γαρίδες που εξειδικεύονται και πρέπει να απασχοληθούμε με αυτούς στα πλαίσια της πολιτικής αλίας. Χαίρομαι γιατί αναφέρθηκε ότι οι αλληλείς, ιδιαίτερα στην Γερμανία, πρέπει να δουλεύουν με πολύ παλαιά σκάφη. Και τώρα, και γίνομαι λίγο πολεμική, εδώ και χρόνια πολλούσαν στις δύο μεγάλες Ολλανδικές εταιρείες και δεν είχαν πια δικές τους οργανώσεις παραγωγών, αλλά ήταν αλυσοδεμένοι όμοιροι αυτών των δύο Ολλανδικών εταιριών, εις ό,τι αφορά τη διαμόρφωση τιμών. Και σωστά το αναφέρατε αυτό. Γι' αυτό έγινε μια μεγάλη απεργία 8 εβδομάδες. Σήμερα τελείωσε η απεργία και με το εμπόριο επετεύχθη μια συμφωνία ώστε να πληρώνουν 3 ευρώ το κιλό. Τώρα, για το καθάρισμα, και αυτό είναι ε, σκάνδαλο, αλλά εύκολα εξηγείται. Πριν από το Μαρόκο ε, πήγαιναν στην Πολωνία και είχε να κάνει αυτό με το ύψος των μισθών. Στο Σλέσβι Χολστάιν δεν υπάρχει κανείς που θα δουλέψει ε, για 3 και 5 ευρώ την ώρα. Κατανοητό. Στο Μαρόκο γίνεται, το δέχονται. Παλιά δέχονταν στην Πολωνία. Ήταν χαμηλή μισθή, τα, τα δέχονταν και ε, ήταν και ευχαριστημένοι. Στο Σλέσβιχ Χόλσταϊν στη Γερμανία και ιδιαίτερα στη Βόρεια Γερμανία, στην ε, Δανία, στην Ολλανδία δεν μπορεί κανείς να ζήσει χωρίς γαρίδες. Όλοι τρελαινόμαστε για αυτές αλλά συχαινόμαστε τα συντηρητικά. Και ένας ε, πραγματικός κατ του Σλέσβι Χόλσταϊν θα πάει στην Τράτα, στην Ψαρόσκαλα και θα αγοράσει επιτόπου τη γαρίδα. Αυτό όμω δεν το μπορούν να το κάνουν όλοι. Και γι' αυτό, όπω και η κυρία Λεβίν, έχω και εγώ το πρόβλημα ότι... Ε, ε, είναι πολύ κονσερβαρισμένες οι κονσέρβες, πολλά προϊόντα τέτοια. Έχει να κάνει αυτό και με το μεγάλο ταξίδι, γιατί θα πρέπει να πάνε στο Μαρόκο και μετά να γυρίσουν και ναι, αφού γίνει η επεξεργασία είναι πολύ μεγάλο το ταξίδι και γι' αυτό ε, είναι και δύσκολο να αποφύγουμε τα συντηρητικά. Όμως αυτό θα πρέπει να το δούμε ως μια τελικά και ενδεχομένως ε, θα πρέπει να αλλάξει η ε, τιμή να είναι κάτι ιδιαίτερο δηλαδή η γαρίδα στο πιάτο μας όταν δεν θα έχει συντηρητικά. Τώρα για τις απορρίψεις, ε, στις συζητήσεις που έκανα με τους αλληλείς Γαρίδας, είπαν ότι θέλουν υποστήριξη για την αναδιαμόρφωση των αλλιευτικών σκαφών και των αλλιευτικών εργαλείων, γιατί λένε ότι μόνοι τους δεν μπορούν να χρηματοδοτήσουν αυτό το εγχείρημα. Τώρα μιλάω για τους Γερμανούς αλληλείς Γαρίδας. Και αν δούμε αυτά τα σκάφη που είναι πια 30 ετών και πάνω, ε, πράγματι θα συμφωνήσουμε μαζί τους. Δεν έχουν τα έσοδα και τα κέρδη που χρειάζονται για να κάνουν επανεξοπλισμό των σκαφών. Εμείς βέβαια δεν είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό. Πρέπει να το πούμε αυτό, εκτός και αν έχω λάθος ενημέρωση, εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τους αλληλείς γαρίδας που ε, δραστηριοποιούνται στη μεικτή αλία. Τώρα για τη μέγιστη απόδοση. Ε, όλοι είναι διατεθειμένοι να... Α, ε, για τις άδειε ε, όλοι είναι διατεθειμένοι να περάσουν από τη διαδικασία, αλλά μέχρι να γίνει αυτό θα τελειώσει και το 2012. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη μελέτη, διότι ε, είναι χρησιμότατη στη δική μου εκλογική περιφέρεια και χαίρομαι πολύ διότι οι Ολλανδοί και Δανείοι συνάδελφοι ε, έχουν έτσι μια πολύ καλή βάση για να δουλέψουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους εισηγητές. Ευχαριστώ, κύριε Γκόρμπατσικ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την παρουσίαση η οποία ήταν ενημερωτικότατη σε ό,τι αφορά την κατάσταση αγοράς και όλο τον τομέα της γαρίδας. Και βεβαίως αυτά ισχύουν και στην Βαλτική που είναι κλειστή θάλασσα και η κυρία Ρόντες είπε επίσης ότι επηρεάστηκε και η παραγωγή. Τώρα έχει αλλάξει λίγο πάλι η κατάσταση εις ό,τι αφορά την, ε, τις αμοιβέ. Υπάρχουν όμως και κάποιες δυνατότητες που ανοίγονται εδώ και πάνω σε αυτό θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση, αυτό που είπατε για τον ε, προϋπολογισμό, τις τιμές μάλλον και τα περιθώρια κέρδους την τιμή ανά που έχουν αυτά τα προϊόντα. Κράτησα το νούμερο 3,5 ευρώ ανά κιλό γαρίδας. Καθαρισμένης γαρίδας. Αυτό είναι η τιμή για τον Αλιέα. 1,55 ευρώ είπατε τιμή στην αγορά είναι πολύ κάτω από το κόστος αν θέλουν οι παραγωγοί να αγοράσουν και καμιά φορά γι' αυτό ξεσπούν απεργίες και υπάρχει αναστάτωση στην, στον τομέα. Σε σχέση με αυτά που είπατε εσείς, ε, που είπατε για αυτή την αρχή υπεύθυνη για τον, την τον ανταγωνιστικότητα, τον ανταγωνισμό και την προστασία των παραγωγών. Δεν θα μπορούσαν δηλαδή να προβλέψουν ε, τιμές ελάχιστες για αυτά τα προϊόντα, γιατί η κατάσταση στην αγορά δεν είναι βιώσιμη. Έχουμε μια κοινή αλληλευτική πολιτική που εφαρμόζεται, έχουμε παγκόσμια πρότυπα που επίσης εφαρμόζονται και πολλές άλλες ρυθμίσεις και κανονισμούς που ε, διέπουν την αλλία. Θα μπορούσαμε λοιπόν να δούμε και αυτό το θέμα της ανταγωνιστικότητας που, στο οποίο πρέπει να δοθεί προτεραιότητα. Επίσης στο Μαρόκο πράγματι η μισθή και η ημερομίσθια είναι πολύ χαμηλότερα τώρα από ό,τι ήταν παλιότερα στην Πολωνία όπου ασχολούνταν και δραστηριοποιούνταν εκεί οι συμπατριώτες μου. Ε, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω μια αναφορά και στην ε, ζάχαρη που είναι το κατεξοχήν παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί όταν πρόκειται για την προστασία των πελατών επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να αγοράζει φθηνή ζάχαρη ε, από άλλες χώρες, τρίτες χώρες και τώρα έχει αυξηθεί κατά 100% η τιμή της ζάχαρης στη χώρα μου. Από μισό ευρώ, α, τώρα πλησιάζομαι για ένα κιλό ζάχαρη το 1,5 ευρώ περίπου. Αυτό δεν ε, ε την ανταγωνιστικότητα δεν, δεν έλαβε υπόψη την ανταγωνιστικότητα, οδήγησε σε κατάρρευση των ε, ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υπέρ των ε, επιχειρήσεων των τρίτων χωρών, με τεράστια αύξηση της τιμής. Αυτό λοιπόν θέλω να το τονίσω, γιατί ε, καλό είναι να μας προβληματίσει και σε σχέση με το τι παθαίνει ένας κλάδος ε, όταν δεχόμαστε πολλές υποχωρήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει ε, και σε άλλους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα για τα, τις απορρίψεις, και αυτό είναι ένα δύσκολο θέμα. 75% λέτε ε, ότι ρίπτονται στη θάλασσα. Περίπου 80%, 80 πολλές φορές. Πολλά ψάρια πεθαίνουν έτσι. Καλό θα είναι λοιπόν να γίνει μια μελέτη για την επιλεξιμότητα για να μειώσουμε τις απορρίψεις ε, υπήρχε μια ε, επιτροπή που εξέτασε το θέμα και είπε ότι θα μπορούσαμε να ε, έχουμε αλλιευτικά εργαλεία που θα επιτρέπουν στα μικρά ψάρια να ξεφεύγουν από τα δίχτυα να ξε, ξεγλιστρούν από τα μάτια. Αυτό στη... Φαίνεται ότι στην περίπτωση της γαρίδας δεν μπορεί εύκολα να γίνει. Δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τέτοια διαφοροποίηση των ματιών για αυτή την επιλεξιμότητα που γίνεται σε άλλα είδη. Άρα λοιπόν δεν θα ήταν καλύτερο να κάνουμε κάποιες έρευνες ούτως ώστε αυτό το 78% ε, των απορρίψεων να το εκμεταλλευτούμε, να το διατηρήσουμε δηλαδή αυτό το, αυτά τα αλλιεύματα και να δούμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε και άλλους ε, ε, κλάδους σε, πολλού, σε πολλές χώρες οι γαρίδες δεν είναι τόσο δημοφιλείς και λόγω της τιμής. Θα μπορούσαμε να το συσκευάζουμε με διαφορετικό τρόπο και πιο οικονομικό τρόπο ίσως και θα μπορούσαμε να δούμε έτσι λίγο από κάποια απόσταση το θέμα αυτό, να συμπεριλάβουμε περισσότερα προϊόντα και να τα κάνουμε πιο δημοφιλή σε ορισμένε χώρες δεν τρώνε καθόλου τι γαρίδε. Ε, καμιά φορά δεν τις γνωρίζουν, δεν γνωρίζουν το προϊόν ή δεν του δόθηκε η ευκαιρία να το δοκιμάσουν γιατί ε, το πετούν. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια ορθολογική προσέγγιση. Δεν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό το προϊόν για να επιφέρουμε κάποιες αλλαγές. Ευχαριστώ κύριε Ραβερτσίκ. Θα ήθελε κανείς άλλος να λάβει το λόγο. Όχι. Καλώς. Θα ακούσουμε τον κύριο Αβιάτρα να απαντήσει πολύ σύντομα στις πολυάριθμες ερωτήσεις που του τέθησαν και ελπίζω να το κάνει με πολύ συνοπτικό τρόπο. Ναι, θα προσπαθήσω ε, να το κάνω συνοπτικά διότι αυτό με υποχρεώνει να κάνω και η απουσία του Τόμας Μπέικερ, διότι εκείνος θα απαντούσε σε όλα αυτά τα θέματα σχετικά με τον εξοπλισμό, τις απορρίψεις κλπ. Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα αφορούσε στις απορρίψεις. Ε, πώς γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πάνω από 82.000 τόνοι. Κοιτάξτε, πρόκειται για μια πολύ λεπτομερή έρευνα από το Ινστιτούτο του Αμβούργου με επικεφαλής του Τόμας Νόιντεκερ και που κατέληξε σε αυτές τις διαπιστώσεις ότι αλλιεύονται 182.000 τόνοι συνολικά. Αυτό που μπορώ να απαντήσω λοιπόν στον πρώτο ερωτώντα είναι ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 τόνοι που επιβιώνουν, 100.000 τόνοι ε, ψαριών που επιβιώνουν. Οι απορρίψεις ή το υπεραλίευμα αφορά σε μικρές γαρίδες ή επίπεδα μικρά ψάρια ε, και άλλα είδη Τώρα, η αυθονία της γαρίδας ε, είναι προφανής, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ψάρι το οποίο να είναι θηρευτής της γαρίδας. Ένα άλλο στοιχείο είναι η υπερθέρμανση των υδάτων στον Βορρά, κάτι το οποίο συνέβαλε στο να φύγουν ακριβώς οι θηρευτές γαρίδας από τις περιοχές αυτές. Ε, σχετικά με το TAC, ε, όταν είπα τάκ και τάξ στον πληθυντικό, δεν εννοούσα τον φόρο, αλλά τα total allowed catch που είναι τα συνολικά επιτρεπόμενα ε, αλλιεύματα. Τώρα, οι αποστολές στο Μαρόκο γίνονται με φορτηγά, όχι αεροπορικός και συνεπώς οι επιπτώσεις ως προς την ποιότητα είναι πιο περιορισμένες. Και υπάρχει μια θηγατρική η οποία είναι εξειδικευμένη στη μεταφορά των ηχθείων. Μια άλλη ερώτηση σχετικά με την ελάχιστη τιμή. Αναφέρθηκα στην ελάχιστη τιμή επί μακρόν και αναφέρθηκα επίσης και στην δικαστική διαδικασία που έγινε από πλευράς ΕΝΕΜΑ της Ολλανδικής Αρχής Ανταγωνισμού ως προς τις ελάχιστες τιμές. Και νομίζω ότι και η κυρία Ροντούστα απάντησε στο ερώτημα. Ελέγχθη ότι πρόσφατα υπήρξε μία συμφωνία σε μια τιμή τριών ευρώ. Και με αυτόν τον τρόπο, με τον πιο απλό τρόπο και βιώσιμο τρόπο, καταπολεμάται και το dumping. Είναι δηλαδή καρπός της ε, συνεννόησης μεταξύ των παραγωγών και των μεταποιητών. Πρέπει να έχω ξεχάσει κάποιες ερωτήσεις, λέει ο μιλητής. Oui, il y avait une question. Oui, on, on, euh, un intervenant a aussi parlé de la... Α, ναι. Ε, κάποιος αναφέρθηκε στη Βαλτική. Πρέπει να σας πω ότι η γκρίζα γαρίδα αλλιεύεται στη Βόρεια Θάλασσα και όχι στη Βαλτική. Ευχαριστώ κύριε Βιάτα. Λυπούμαστε που δεν είναι εδώ ο κύριος Νόιντεκερ ο οποίος θα ήταν σε θέση να απαντήσει λεπτομερέστερα σε ερωτήσεις. φαίνεται ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια να ενταχθεί η Ισλανδία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον η τέφρα της Ισλανδίας. Συγγνώμη, ήταν ε, αστιάκι αυτό που έκανα. Και περνούμε τώρα στο επόμενο σημείο. Σας ευχαριστούμε ακόμη μια φορά κύριε Βιάτ. Και περνούμε στο επόμενο σημείο λοιπόν. Πρόκειται για την παρουσίαση ενός ενημερωτικού σημειώματος σχετικά με τη βιομηχανική αλληλεία στην Βαλτική θάλασσα. Ο κύριος Hans Lassen που είναι ε, ανεξάρτητος εμπειρογνώμων, πρώην διευθυντής της CM, δηλαδή της, ε, του Διεθνού Συμβουλίου ε, εκμετάλλευσης των θαλασσίων πόρων. Υπάρχει λοιπόν μια σύντομη μελέτη και η οποία είναι στη διάθεσή σας στα αγγλικά, γερμανικά, πολωνικά και σουηδικά. Ε, και πρόκειται για την παραγωγή ηχθιαλεύρων και ηχθιελαίου από σαρδελόρεγγες και ρέγγες. Κυρίες και κύριοι, αν θέλετε θα δώσω αμέσω το λόγο στον κύριο Λάσεν, ο οποίος θα μας κάνει την παρουσίαση. Κύριε Λάσεν, έχετε περίπου 20 λεπτά στη διάθεσή σας για την παρουσίαση αυτή. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ που με καλέσατε να κάνω αυτή τη σύντομη παρουσίαση για τη βιομηχανική αλληλεία στη Βαλτική. Όταν μιλάμε για βιομηχανική αλληλεία στη Βαλτική, μιλάμε για σαρδελόρεγγα και ρέγγα. Επανέρχομαι σε αυτό που εννοούμε με τα συστατικά, τι είδους δηλαδή συγκεκριμένα ρέγγα, σαρδελόρεγγα, πάντως για αυτά τα δύο είδη μιλάμε. Το βασικό κομμάτι της αλίας αυτής λαμβάνει χώρα ε, στην ανατολική περιοχή της Βαλτικής. Θα δώσω και αργότερα λεπτομέρειες. Τέλος, τελευταία και παρατήρηση, χρησιμοποιούμε δύο βασικές χρήσεις των βιομηχανικών αλλιευμάτων, ας πούμε. Είναι η χθιάλευρα και η χθιέλεα πρώτον, και το άλλο είναι ζωοτροφές. Τώρα, ποια είναι τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται και πάω στην αγορά ηχθιελέ, ηχθιαλεύρων και ηχθιελαίων. Μαζί πάει αυτό. Πάμε, ε, ε, ε, χρησιμοποιούνται στην ε, υδατοκαλλιέργεια και το ποσοστό ε, υπάρχει ενδεικτικά, αντικατοπτρίζει την παγκόσμια αγορά. Η, αγορά της ε, ηχθιοκαλλιέργειας είναι εδώ η κυρίαρχη. Αν προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα βιομηχανικά λιεύματα, πρέπει να δούμε τα σημεία εκφόρτωσης, ε, την εκφόρτωση που πάει απευθείας στην ανθρώπινη κατανάλωση ή νοπά ή μεταποιημένα, μαριναρισμένα ή οτιδήποτε άλλο. Ε, η επεξεργασία γίνεται στη Δανία κυρίως εδώ για να πάνε για ηχθιάλευρα και ζωοτροφές και υπάρχουν και άλλα τα οποία πάνε κατευθείαν ε, ως νοπά ή άλευρα και έλαια για ζωοτροφές. Τώρα, δεν υπάρχουν ε, άμεσα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία για τον άμεσο αριθμό της παραγωγής. Ε, μιλάμε για περίπου 300.000 τόνους ετησίως που είναι μια αξία περίπου μεικτά 30 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ένα θέμα που ανέφερα ήδη εισαγωγικά είναι ότι μιλάμε για ρέγγα και σαρδελόρεγγα εδώ και παρουσιάζω κάποια δείγματα που υποδεικνύουν ότι όλα αυτά τα λιεύματα πράγματι ε, είναι σαρδελόρεγγα και ως ένα βαθμό αλλά ο μπακαλιάρος ε, είναι ελάχιστα μεταξύ των αλλιευμάτων. Δεν έχουμε δηλαδή μεγάλο πρόβλημα παρε, παρεμπιπτών των αλλιευμάτων εδώ. Είναι κυρίως Λερέγκα και Σαρτελόρεγκα. Σε αυτή τη γραφική παράσταση βλέπουμε λίγο και τα αλλιευτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται. Είναι τράτες, ε, τράτες βυθού, ε, υπάρχει επαφή δηλαδή, ε, υπάρχει μικρό άνοιγμα ε, ματιών, υπάρχουν κανονισμοί που το, τα περιορίζουν στα 16 χιλιοστά και αν δείτε τον αλλιευτικό εξοπλισμό θα δείτε ότι είναι 16 22 χιλιοστά το χαρακτηριστικό άνοιγμα που χρησιμοποιείται. Τώρα για τη ρέγγα έχουμε ελάχιστο 32, αλλά οι, οι τράτες είναι περίπου 16-22 χιλιοστά. Looking on the fleets which operates here, ε, Ο κλάδος είναι αρκετά μεγάλος. Δεν μπόρεσα να βρω διεθνή στατιστικά στοιχεία. για τα βιομηχανικά σκάφη. Έχω πάρει τράτες πάνω από 24 μέτρα ως μέτρο μέτρησης και το βασικό μήνυμα από αυτό το γράφημα είναι ότι βλέπουμε μείωση του στόλου των αριθμών των σκαφών. Δηλαδή, αν δούμε με την υποδύναμη, πάλι υπάρχει μείωση, η ίδια τάση. Αυτό αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι ο κλάδος γίνεται πιο αποτελεσματικός ή αποδοτικός καλύτερα τα τελευταία χρόνια και σε αυτό το στόλο όπως και σε άλλους τομείς ε, υπάρχει υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό με την έννοια ότι υπάρχει στόλος που θα μπορούσε να λιεύει περισσότερο από, ε, από τα διαθέσιμα αποθέματα και γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ε, πτωτική τάση τώρα. Μετά συνολικές εκφορτώσεις Πάλι μιλάμε εδώ για τα δύο κύρια είδη ρέγγα, Σαρδελόρεγκα, που είναι από θέματα με σχετικά σταθερές εκφορτώσεις τα τελευταία χρόνια. Είναι περίπου 700.000 τόνοι το σύνολο. Λίγο πάνω από το μισό είναι Σαρδελόρεγκα, έτσι χονδρικά. Δηλαδή είναι 400.000 η Σαρδελόρεγγα, 300.000 η Ρέγγα. Αν δούμε τώρα την παραγωγή ηχθιελαίων και ηχθιαλεύρων, τρία εργοστάσια υπάρχουν ουσιαστικά που κατασκευάζουν αυτά τα ηχθιάλευρα και τα ηχθιέλεα με πρώτη ύλη από αυτά τα ψάρια στη Δανία. Ε, δύο είναι σε λιμάνια στο Σκαγεράκι ή στη Βόρεια Θάλασσα. Το ένα που είναι προς τον Σκαγεράκι είναι στα όρια μεταξύ Σκαγεράκι και Βόρεια Θάλασσα. Οι δύο μεγάλες χώρες που δίνουν την πρώτη ύλη για αυτή την παραγωγή είναι η Δανία και η Σουηδία, αλλά αν δούμε τα στατιστικά οι περισσότερες από τις άλλες χώρες της Βαλτικής δίνουν και αυτές μικρότερα ποσά πρώτης ύλη τα οποία μεταποιούνται. Η βασική όμως παραγωγή είναι Δανία-Σουηδία. Να επαναλάβω εδώ πάλι ότι δεν μπόρεσα και δεν νομίζω ότι υπάρχουν στατιστικά στοιχεία που θα σας επιτρέψουν να βρείτε συγκεκριμένα τον αριθμό, επακριβή αριθμό των ψαριών που χρησιμοποιούνται από αυτά τα πελαγιακά αποθέματα για ηχθιάλευρα και ηχθιέλευρα. Γιατί ε, υπάρχουν αλλαγές στις στατιστικές μεθόδους από το 2011 και γι' αυτό προς το παρόν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Προσπάθησα να σας δώσω όμως κάποια στατιστικά στοιχεία για την χρήση της παραγωγής των πελαγικών ειδών και πάλι εξαιρώ την Δανία όταν μιλάμε για τον κλάδο γιατί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των προϊόντων των Δανέζικων έρχονται από τη Βόρεια Θάλασσα. Υπάρχουν τεχνικά μέτρα που ισχύουν για την βιομηχανική αλία στην Παλτική. Τα συνοψίζω εδώ, τα πήρα από τον κανονισμό. Καταρχήν υπάρχει κανονισμός για τα παραλιεύματα, ε, που δεν επιτρέπεται πάνω από 3% ε, μπακαλιάρος και ανάλογα από το είδος στόχο προβλέπονται τα χιλιοστά. Θα πρέπει δηλαδή να στοχεύσετε στα 16 χιλιοστά για την Σαρδελόρεγγα και Ε, στον βορρά χρησιμοποιείται, χρησιμοποιούνται και εξοπλισμοί για μικρή ρέγγα. Για την ρέγγα είναι λίγο διαφορετικά τα δεδομένα σε σχέση με την σαρδελόρεγγα. Ε, και τα μεγέθη τους διαφοροποιούνται. Ε, κυρίως ε, το, το βασικό αλλιευόμενο προϊόν είναι η σαρδελόρεγγα ε, στη, στο κέντρο, στην κεντρική Βαλτική. Τώρα, τα ΤΑΚ για το 2011, η γενική τάση είναι για τη Ρέγγα και τη Σαρδελόρεγγα ε, σημειώθηκε μείωση στα ΤΑΚ για το 2011, συνολικά επιτρεπόμενα ε, αλλιεύματα σε σχέση με το 2010, γιατί αυτό αντικατοπτρίζει τη μείωση στα αποθέματα. Θα επανέλθω όμως λίγο αργότερα στο θέμα αυτό για να το δούμε ε, μέσα σε ένα μακρότερο χρονικό ορίζοντα. Καταρχήν για τη Σαρδελόρεγγα έχουμε από θέματα όπου η θνησιμότητα των ηχθείων αυξήθηκε Είμαστε σε ένα επίπεδο ε, το οποίο είναι επικίνδυνο αν λάβουμε υπόψη μας τη μέγιστη διαρκή απόδοση. Βέβαια δεν είναι επικίνδυνα, ε, επικίνδυνες οι ενδείξεις, δηλαδή η υψηλή θνησιμότητα των ψαριών δεν είναι επικίνδυνο σημάδι, απλώς είναι ενδεικτικό. Η σαρδελόρεγγα είναι δύσκολο είδος όμως, γιατί παρουσιάζεται διακύμανση στην ανανέωση του αποθέματος ε, μέσα από την είσοδο νέων ψαριών δηλαδή. Εδώ το δείχνουμε αυτό, δεξιά, ανανέωση δηλαδή. Ευτυχώς είναι υψηλή ε, η ποσότητα των νεαρών ψαριών της Σαρντελόρεγκας που εισέρχονται στο απόθεμα. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο απόθεμα για τη Ρέγκα στη θάλασσα Μπόθνια. Εδώ μιλάμε για φιλανδική αλία. Εδώ είναι ε, υψηλό το απόθεμα η αναπαραγωγή είναι καλή. Βλέπετε κάτω δεξιά αυξάνονται τα αποθέματα από το 80 μέχρι την αρχή της δεκαετίας του 90 αυξάνονταν και παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα. Η θνησιμότητα των ηχθείων είναι κάτω από το επίπεδο της μέγιστης διαρκούς απόδοσης και τα ε, ε, θέματα είναι υψηλά και η ε, βιομάζα αναπαραγωγής. Οπότε δεν υπάρχουν από εκεί κίνδυνοι. Υπάρχουν βέβαια και, άλλες, ε, και άλλα αποθέματα ρέγγας στη Βαλτική. Υπάρχουν παρόμοια γραφήματα που θα τα βρείτε στην έκθεση, αλλά αυτά λίγο συμβάλλουν μόνο στη βιομηχανική αλληλεία και δεν είναι άμεσα ο στόχος αυτός των αποθεμάτων. Συνοψίζω. Οι προοπτικές για τη Σαρδελόρεγγα είναι σχετικά ε, καλές. Όταν θέλουμε να αποτιμήσουμε την κατάσταση στη Βαλτική πρέπει να θυμόμαστε ότι τα αποθέματα στη Βαλτική σε σχέση με τη Βόρεια Θάλασσα ή άλλα αποθέματα επηρεάζονται περισσότερο από τις περιβαλλοντικές αλλαγές και τις διακυμάνσεις από τι άλλα αποθέματα ηχθείων και γι' αυτό στοχεύομαι στο να κρατήσουμε την θνησιμότητα των ηχθείων έλεγχο, ενώ η διακύμανση της βιομάζας δεν είναι τόσο σημαντική γιατί είναι αναπόφευκτη σε ένα σύστημα όπως αυτό της βαλτικής, ε, τη βιομάζα αναπαραγωγής δηλαδή, που διαφοροποιείται. Γιατί ε, τα πελάγια είδη στη Βαλτική διαφέρουν και πολλά πελάγια είδη διαφέρουν από, στη Βαλτική σε σχέση με άλλα. Τέλος, Η Βαλτική και τα αποθέματά της υποφέρουν από διοξίνες, υψηλή συγκέντρωση διοξινών, που δεν περιορίζεται μόνο στα πελάγια είδη, αλλά και τα πελάγια είδη παρουσιάζουν αυτό το φαινόμενο. Και θα πρέπει αυτό να το λάβουμε υπόψη μας όταν ε, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τους διαθέσιμους πόρους είναι δυνατόν από τεχνολογικής πλευράς να φτιάξουμε ηχθιάλευρα και ηχθιέλεα, τα οποία να τηρούν την προβλεπόμενη νομοθεσία εις ό,τι αφορά τις διοξίνες και τα PCB, τα πολυχλωριωμένα διφενήλια. Άρα λοιπόν, ποια είναι τα βασικά μας ευρήματα. Καταρχήν έχουμε ένα σύστημα καλά τεκμηριωμένο. Υπάρχουν πολλά στατιστικά στοιχεία για τα ψάρια αυτά. Έχει γίνει αποτίμηση των αποθεμάτων. Ε, είναι λίγες οι απορρίψεις εδώ. Η αλία, η παράνομη, λαθρέα και άνερχη, άναρχη δεν έχει το τεκμηριωθεί ως μείζον πρόβλημα. Υπάρχουν παραδείγματα εδώ με βραχίες περιόδους κάποιων προβλημάτων ε, με κάποιους αλληλείς, αλλά τέλος πάντων αυτό δεν συνιστά μεγάλο πρόβλημα λαθραλίας εδώ. Οι στόλοι μειώνονται, το είπαμε αυτό, οι τάσεις ε, στα αποθέματα διαφοροποιούνται, δεν είναι ομοιόμορφες. Υπάρχει διαφορετική διακύμανση μεταξύ των αποθεμάτων, υπάρχουν περιβαλλοντικές επιδράσεις που είναι διαφορετικά. Δεν είναι το συγκεκριμένο είδος η, η αλίευσή του που επηρεάζει την διακύμανση. Πίεση τώρα εκμετάλλευσης. Είναι λίγο πάνω από το στόχο του MSY, μέγιστη διαρκούς απόδοσης. Όταν μιλάμε για σαρδελό και ένα απόθεμα ρέγγας, η βιομηχανική αλία εδώ είναι η βασική αλλιευτική συνιστόσα και γι' αυτό επηρεάζει η βιομηχανική αλληλεία τα αποθέματα ιδιαίτερα γι' αυτό το λόγο κυμαίνεται το απόθεμα Σαρδελόρεγκας. Ας δούμε τώρα λίγο την αγορά. Φαίνεται ότι οι τιμές για την ανθρώπινη κατανάλωση είναι σημαντικά υψηλότερες από ότι για τη βιομηχανική χρήση των αλλιευμάτων. Αλλά σε ορισμένες περιοχές είναι πολύ μικρή η ανθρώπινη κατανάλωση για τη σαρδελόρεγγα στη Δανία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία. Ε, είναι πολύ... Δεν φαίνεται ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη κατανάλωση πολύ. Αλλά υπάρχει στην Ανατολική Ευρώπη. Αυτά εν συντομία για τη βιομηχανική αλία στη Βαλτική. Να σημειώσω ένα τελευταίο ότι η βιομηχανική αλληλεία σε αντιπαράθεση με τη Βόρεια Θάλασσα δεν υπόκειται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα κανονιστικό πλαίσιο. Εδώ, για αυτή την αλληλεία, έχουμε ένα κανονιστικό πλαίσιο ανεξάρτητο χρήσης. Ελπίζω να τα είπα όλα αυτά που έπρεπε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, the picture on the left hand side is from Helsinki. Α, και ο κύριος, ε, έχουμε και τον κύριο από... Α, στο ε, Ελσίνκι θα γίνει ένα φεστιβάλ Ρέγκας και έχουμε εκπρόσωπο. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια να δώσουμε το λόγο στους συναδέλφους που ζήτησαν το λόγο. Πρώτος ο κύριος Λοντότσικ. Dziękuję bardzo. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εγώ... Για να δούμε. Τώρα που το πιάσαμε επιτέλους αυτό το θέμα, γιατί μας πήρε πολύ χρόνο, αλλά τώρα φτάσαμε σε αυτό το σημείο και θα πρέπει να εκφράσουμε ευχαριστίες. Γιατί πράγματι ανοίξαμε το θέμα αυτό. Αναφέρομαι σε μία δήλωσή σας που τη θεωρώ αμφιλεγόμενη γιατί είπατε ότι οι προοπτικές φαίνονται να είναι καλές. Ενώ εγώ κατάλαβα ότι αυτά που είπατε δείχνουν σαφώς ότι οι προοπτικές δεν είναι καλές. Και όλα αυτά που μας είπατε δείχνουν ότι Δεν πρέπει κανείς να εκπλήσεται, στη Δανία για παράδειγμα, δεν πρέπει ο κόσμος να εκπλήσεται ε, από την ε, αντιμετώπιση του θέματος. Να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Σε σχέση με τα συμπεράσματα, αν κάποιος δεν είναι ειδικός μπορεί και να συμφωνούσε για τα στοιχεία, για τα αποθέματα, για το στόλο, παρουσιάζεται εδώ τεκμηρίωση, επίσης και οι πόροι φαίνονται να είναι εντάξει, τα αλλιεύματα σε καλό επίπεδο, ότι φαίνονται όλα αυτά ωραία από τις στατιστικές. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε πάρει πληροφορίες ε, από την Κομισιόν που μας ενημερώνει ότι δεν ξέρει τι γίνεται στη με, τη Ρέγκα, ούτε οι επιστήμονες. Εσείς μας είπατε ε, ότι είναι 400.000 οι τόνοι της Ρέγκας και ακόμα δεν ξέρουμε πώς θα τι επιπτώσεις θα έχει όλη αυτή η αλίευση στη Βαλτική. Διότι η Βαλτική έχει ιδιαιτερότητες και είναι και υποπροστασία σε μεγάλο βαθμό. Ακούγεται ηρωνικό, αλλά επηρεάζονται ε, και άλλα είδη. Γιατί ακριβώς λόγω της ιδιαιτερότητας της Βαλτικής. Βέβαια, ε, ε, φαίνεται ότι είναι σημαντικά αυτά τα δύο, ε, Ρέγκα Σαρτελόρεγκα, αλλά και άλλα ήδη έχουν πρόβλημα. Και σε άλλα σημεία δεν μπορώ να συμφωνήσω μαζί σας. Τώρα, και για το γάδο και για άλλα ψάρια. Ε, δεν έχουν γίνει έρευνες. Είπατε ότι διεξάγονται τώρα, αλλά γιατί για το στόλο, ας πούμε, δεν έχουν γίνει μελέτες για τις επιπτώσεις ε, των εξελίξεων. Είπατε ότι υπάρχει και στατιστικό πρόβλημα με τα λιεύματα και αναφέρεται και αυτό επίση στη σελίδα 24 του εγγράφου σας που λέτε ή κάπου πάντων λέτε ότι τα δανέζικα λιμάνια δεν καταχωρούν πολλά στοιχεία δηλαδή πολλά θέματα παραγνωρίζονται Οπότε γίνονται εκφορτώσεις ως έτυχε σε μεγάλο βαθμό. Δεν ξέρω, ε, θα πρέπει να προσδιορίσουμε τι ακριβώς προέρχεται από τη Βαλτική. Ίσως γι' αυτό να έχουμε και το μεγάλο πρόβλημα. Γι' ε, αυτό να μειώνονται και τα αποθέματα στο τέλος. Επίσης, ε, παραγωγή ηχθιαλεύρων και ηχθιελαίων. μας είπατε για την παραγωγή. 400, λέτε ακόμα περίπου 400.000 και ίσως ε, αν συνεχίσει να είναι χαλαρός ο έλεγχος θα μας πάρει χρόνια μέχρι να καταλάβουμε τι γίνεται ακριβώς. Θα πρέπει συνέχεια να προσαρμόζουμε το σύστημα ώστε να παίρνουμε τα στοιχεία που θέλουμε κάθε φορά γιατί τα υπάρχονται δεν επαρκούν. Επίσης θα ήθελα να πω Κάτι ακόμα. Λέει στο κείμενό σας ότι ε, υπάρχουν συγκρίσεις μεταξύ αλλιές για ανθρώπινη κατανάλωση και για ζωοτροφές. Δεν μπορώ να συμφωνήσω εδώ. Ε, ε, αναφέρονται η Σουηδία και η Δανία που δεν τρώνε ε, ρέγγα και σαραδελό ρέγγα σχεδόν καθόλου. Άρα όλη η ποσότητα πάει στο βιομηχανικό τομέα για να γίνει ζωοτροφή. Δεν μπορώ λοιπόν να μιλήσω για ε, σύγκριση στην κατανάλωση αφού κατανάλωση δεν υπάρχει. Επίσης μιλήσατε για ένα άλλο θέμα, ότι ας πούμε είναι κλειστή θάλασσα. Ε, υπάρχουν διαφορετικές περιοχές, Μπόθνια ε, ε, και άλλες, με διαφορετικό βάθος. Είπατε ότι δεν επηρεάζεται η βιομηχανική αλληλεία, δεν διαφοροποιεί. Τώρα αυτά τα παρασυρώμενα δίχτυα τι κάνουν. Έχουμε δεδομένα έχουμε ελέγχους 150 δειγματοδηληπτικοί έλεγχοι έγιναν ε, πέρσι σε ποσότητα εκφόρτωσης περίπου 100.000. χωρίς επακριβή διαφοροποίηση ειδών. Τα δεδομένα από την 1η Πρώτου του 2011 στηρίζονται στους υποχρεωτικούς ελέγχους και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας είπε πόσο σημαντική είναι η έλεγχη και για τη ζωοτροφή, δηλαδή τα προϊόντα που θα πάνε για ζωοτροφή. Ε, ε, είναι ελάχιστα τα επιστημονικά δεδομένα. Ε, επίσης κάτι άλλο, οι λανθασμένες πληροφορίες, τα σφάλματα και στα έγγραφα και στα βιβλία, τα ημερολόγια των πλοίων σχετικά με τα αλλιεύματα. Λένε ότι οι αλληλείς δίνουν τα δεδομένα, αλλά πώς ε, αξιολογούνται. Πολλές φορές γίνεται σύγχυση μεταξύ ε, ε, σαρδελόρεγκας και ρέγκας. με αποτέλεσμα να ε, δίνονται λάθος σημεία και να μειώνεται ο, να φαίνεται ότι μειώνεται ο ε, πληθυσμός της Ρέγκας. Επίσης, ε, τα προηγούμενα χρόνια ακούμε ότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δεν έγιναν. Τώρα άρχισαν να γίνονται. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και η Ιζαμπέλα ε, μίλησε και για την ε, άναρχη παράνομη λαθρέα αλία. Και εκεί γίνεται ε, παράνομη αλία και το, τα παράνομα κέρδη είναι κάτω κάποια εκατομμύρια ευρώ. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε τον κίνδυνο. Πόσο μεγάλη είναι η απειλή. Επίσης, Ε, θα επηρεαστούν και ο γάδος, ο μπακαλιάρος ε, πέρα από την, ε, μετά από την Ρέγκα και την Σαρδελόρεγκα. νομίζω ότι είναι εσφαλμένη η εκτίμηση ότι μειώνονται τα αποθέματα γάδου. Τελευταία ερώτηση. Προσοχή όταν μιλάμε για τις απορρίψεις ε, στα πλαίσια της βιομηχανικής ελίας, γιατί όλα τα πετάνε μέσα στο μηχάνημα και μετά τα αλέθουν εκεί, τα συσκευάζουν και μετά ε, γίνονται ζωοτροφές. Συγγνώμη που τα είπα έτσι με συναισθηματική φόρτιση, αλλά είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα κέριο ζήτημα αυτό για μένα και με ενοχλεί που γίνεται σύγχυση μεταξύ των θεμάτων και δεν ακριβολογούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια για την εισήγηση. Πραγματικά χρειαζόταν κάτι τέτοιο. Όσον αφορά το τι γίνεται με τους πόρους στα πελαγικά ήδη. Έχω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Υπάρχει τίποτα το κατάλαβα την παρουσίαση. Πέστε μου τα εξής όσον αφορά το συνολικό αλίευμα των πελαγικών για όλες τις βαλτικές χώρες. Πόσα από αυτά πάνε για ανθρώπινη κατανάλωση πόσα πάνε για ζώα, πόσα πάνε για μηχανικούς σκοπούς και πόσα πάνε για τους ανθρώπους. Κάτι άλλο τώρα, όσον αφορά τα ηχθιάλευρα και τα ηχθιέλαια. Όπως γνωρίζουμε και όπως γράφει η έκθεση, η Βαλτική θάλασσα και Σαρδελόρεγγα αλλά και η έχουν πάρα πολλές διοξίνες, πάρα πολλά PCB πολλά από αυτά τα είδη πηγαίνουν για τη βιομηχανία, αλλά νομίζω ότι για την, ε, για την ανθρώπινη κατανάλωση πρόκειται για πάρα πολύ ακριβά, ε, πάρα πολύ ανθυγιεινά τρόφιμα λόγω αυτής της συγκέντρωσης του PCB. Όμως, πάρα πολλά από αυτά πάνε για χθιοκαλλιέργεια. Πάνε, ας πούμε, για να ταΐσουν τους σολομούς τη ηθοκαλλιέργειας. Επομένω, τι έλεγχο υπάρχει. Όσον αφορά σε αυτή την ουσία που υπάρχει στα ψάρια για τα οποία μετά πηγαίνουν γίνονται κάλυβρα κλπ. Τώρα, τι γίνεται με τα παραλίευματα του μπακαλάου. Κοιτάξτε, πάρα πολλέ από αυτέ τι ε, τράτες έχουν τεράστια δίκτυα, 30-40 μέτρα. Όμως εκεί πέρα πάμε για σε βάθος 50 μέτρων στην ε, θάλασσα. Ε, άρα πώς θα αποφύγετε την αλίευση του βακαλάου. Ε, καλά συνήθως σε αυτά τα είδη κολυμπάνε στα βαθιά, αλλά τι θα γίνει άμα πάνε πιο πάνω. Πώς θεωρείτε ότι αυτά τα στοιχεία που μας δίνετε είναι αξιόπιστα όσον αφορά το παραλίμμα σε Βακαλάο. Τώρα άλλη μια ερώτηση όσον αφορά τους ε, ε, ψάραδες και το τι πηγαίνει σε ανθρώπινη κατανάλωση σε σχέση με την ρέγγα. Τελικά περισσότεροι περισσότερα πανούνται όσον αφορά τα ψάρια τα οποία πάνε η ανθρώπινη κατανάλωση και γιατί γίνεται παρεσχή αυτό, ότι πάρα πολλά από τα λιέματα πάνε για ζωοτροφές. Και έχουμε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία ε, αυτά τα ψάρια που χρησιμοποιούνται για να τραφούν άλλα ψαριμένως, τι γίνεται με Μιλάμε για τεράστιε ποσότητε που πάνε οι ανθρώπινη κατανάλωση. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο που να, να έχουμε ηχθιάλευρα στα γουρούνια τα οποία τρώμε, στο χοινό που τρώμε και στο κοτόπουλο που τρώμε. Τώρα μια σκέψη γενικού χαρακτήρα παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να εξετάσουμε τι διαφορετικέ χρήσει αυτών των ε, εκφορτώσεων σε, σε κάθε χώρα γιατί κυρίως η Σουηδία και η Δανία ε, αξιοποιούν ε, αυτά τα ελλείμματα για δημιουργημένους χώρους και Λιθουανία, Λετωνία, Πολωνία είναι οι χώρες που χρησιμοποιούν ε, αυτά τα ψάρια για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτό είναι μια παράδοση και είναι και τελικά η προτίμηση του καθενός, η επιλογή του. Όμως Έχουμε επίσης σαρδέλα σαρδελόνικα που τη δίνουμε στους Σολομούς. Αλλού το κάνω αυτό, αλλού όχι. Πάντως, ελπίζω τα PCB να μην υπάρχουν στο τελικό προϊόν που τρώμε. Πάντως είναι σωστό, είναι δεδομένη η υπεραλίευση του βακαλάου. Και έχουμε όλα αυτά τα ψάρια, σαρδέλα, σαρδελόγια που πάνε στους ε, σολομούς και τώρα πάρα πολύ σολομό γιατί μπορούμε να πιάσουμε σαρδέλα, Σαρδελόνικα γιατί, που χρησιμεύουν για την διατροφή του σολομού. Άρα θα πρέπει κανείς να κάτσει και να σκεφτεί τι γίνεται, τι θα γίνει όταν ε, τα αποθέματα ανέβουν του βακαλάου στη Βαλτική, όταν αυξηθούν πάλι όλοι εκείνοι οι οποίοι έχουν ε, επενδύσει σε σκάφη και εξοπλισμό για τα πελαγικά, τι θα γίνει. Θα ψαρεύονται λιγότερο πελαγικά είδη στη Βαλτική και θα συμφέρει περισσότερο να έχει κανείς ε, μικρότερα σκάφη για ε, τα μικρότερα είδη του, της Βαλτικής. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν έχετε νομοθετήσει κάποιο είδου όριο, κάποιο είδου τάκ για ρέγγα, σαρδελόρεγγα. Φαντάζομαι ότι γιατί θα αλλάξουν τα δεδομένα μόλι μπορέσει να ξεφύγει ο βακαλάος από την προστασία του, της μεγίστης ε, επιτρεπόμενης ποσότητας. Να φύγει ο βακαλάο από την διαρκή απόδειξη. Ευχαριστούμε. Ε, πρόεδρο. ευχαριστούμε στην αρχή που σας είπατε ότι έχουμε 400.000 τόνους κάθε χρόνο που πηγαίνουν για χρήσεις μη ανθρώπινης διατροφής, για, για, για, για ζωοτροφή. Πέστε μας πόσο πάνε η πόσο πάνε η τι γίνεται, τελικά τα στοιχεία αυτά αφορούν και, και τις δύο χρήσεις ή για όλο. Επίσης είπαμε ότι έχουμε μόνο τρεις εταιρείε που ασχολούνται με αυτό. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα μητρό των εκφορτώσεων γιατί πέραν αυτού θα, ξέραμε σε αυτά τα τρία εργοστάσια πόσε ζωοτροφές ε, τελικά βγάζουν και τελικά τι γίνεται. Πόσα ψάρια χρησιμοποιούνται για να φτιαχτεί ένα κιλό από ήχθη άλευρο και τέλο πάντων τα ψάρια που πάνε εκεί δεν χρησιμεύουν για τίποτα άλλο. Άρα γι' αυτό είπαμε ότι καταρχήν δεν χρειάζεται έλεγχο παρά μόνο λόγω της ύπαρξης των διοξινών. Για να το δούμε καλύτερα. Ε, ε, μας είπατε δεν υπάρχουν στοιχεία. Και τελικά αυτό μολυνόμεθα. Μια που τρέφουμε τα ζώα με ηχθιάλευρα μολυσμένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη μελέτη. Ευχαριστώ που επιτέλους κάποιος κατάφερε να προκαλέσει τόσο πολύ τον συνάδελφο Ροπατσέκ ε, ώστε να επιδείξει τόσο ταμπεραμέντο. Σοβαρά τώρα να κάνω τις ερωτήσεις μου. Για την ε, υδατοκαλλιέργεια, μια ερώτηση. Η υδατοκαλλιέργεια καταναλώνει ηχθιάλευρα και ηχθιέλαια. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Ένα πρόβλημα είναι το θέμα του λευκόματος, γιατί πρόσφατα πήγα στο Κίελο στο Πανεπιστήμιο που υπάρχει ε, μια, ένα τμήμα που κάνει δοκιμές για τα λευκόματα. Στην υδατοκαλλιέργεια και πώς μπορούν να παραχθούν διαφορετικά. Μακροπρόθεσμα συμφωνείτε, δηλαδή μπορεί να μην κάνουμε τα πολύτιμα ψάρια ηχθιάλευρα και ηχθιέλεα. Επίσης είπατε στην ομιλία σας ότι η Ρέγκα στη Βοθνία ε, είναι υγιής, είναι χαμηλή θνητότητα, δεν υπάρχει κίνδυνος είπατε. Αλλά ταυτόχρονα είπατε ότι άλλα αποθέματα Ρέγκας στην Βαλτική έχουν προβλήματα. Δηλαδή ποια είναι αυτά τα αποθέματα που έχετε υπόψη σα. Είμαστε καλά ενημερωμένοι ότι για παράδειγμα τα αποθέματα ρέγκα στη, στο Μέκλενμπουργκ, Πομερανία, εκεί στις ακτές έχουν πρόβλημα. Και είπατε επίσης ότι η αλλαγή στο περιβάλλον γίνεται όλο και πιο αισθητή. Τι εννοείτε δηλαδή ε, έχει να κάνει αυτό με τα προβλήματα στην Πομερανία Μέκλενμπουργκ. Μπορείτε να μας πείτε λεπτομερέστερα ποια περιβαλλοντικά προβλήματα υπάρχουν και πώς αυτά επιδρούν στα αποθέματα. Γιατί εγώ ξέρω ότι οι ε, σε ορισμένες περιοχές η ρέγγα καταστρέφεται, πεθαίνει, η θνησιμότητα είναι υψηλή. Ευχαριστώ και εγώ για την ομιλία σας. Είναι ενδιαφέρον ότι ένα μεγάλο μέρος των ε, περιοχών αλληλείας ε, ανατολικά της Γρυλανδίας, στη Βαλτική, ε, δεν μας έχουν απασχολήσει με προβλήματα στην Επιτροπή Αλίας παρόλο που υπάρχει η Φιλανδική θάλασσα, η Βόθνια, ε, η ακτή των βαλτικών δημοκρατιών, η Πολωνία από τη μια, μετά η Σουηδία και η Φιλανδία, όλες είναι χώρες ε, που ενδιαφέρονται για τη Βαλτική. Είναι λυπηρό ότι 60.000 ε, τόνοι ρέγγας και σαρδελόρέγγας ε, μεταποιούνται και γίνονται α, δευτερεύουσα σημασίας και μικρής αξίας προϊόντα ενώ για κάθε τόνο τάκ δίνεται σκληρή μάχη για να τα βγάλουν πέρα οι αλλοίς. Το είπε και η κυρία Ρόντες. Η ρέγγα της Βαλτικής στην κατεγά, στο, στον κατεγάτη Σκαγεράκη ε, δεν είναι επαρκή και στη δική μου την ε, περιοχή ε, οι επιστήμονες λένε ότι έπρεπε να μειωθούν ριζικά τα τάκ και το δεχτήκαμε γιατί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα. Σε μια ανατολικότερη ε, θάλασσα που ε, έχει πολύ λιγότερη ανταλλαγή των, και εναλλαγή των υδάτων σε σχέση με τη Βόρεια Θάλασσα ε, τα αποθέματα, οι πληθυσμοί Ρέγκας και Σαρδελόρεγκας εκεί είναι σχετικά σταθερά τα αποθέματα, οι πληθυσμοί σταθεροί. Ε, ο γόνος ε, πώς αναπαράγεται, βρίσκουν τρόφιμα, πώς εξελίσσεται η κατάσταση στις ανατολικότερες περιοχές, στην Πομερανία και στην αλυσίδα της τροφής βλέπουμε ότι ρέγγα σαρδελόρεγγα γίνονται ζωοτροφές μέσα από την ε, ε, ηχθειοκαλλιέργεια περνάνε στην αγορά πάλι τα προϊόντα αυτά. Το 56% των προϊόντων αυτών ε, καταναλώνονται ως τροφή στην ηχθειοκαλλιέργεια και σε ζωοτροφές. Εντάξει, δεν είναι ασύνηθες. Θυμάμαι και από μικρός που τη ρέγγα σε πολύ πιο περιορισμένο βαθμό την χρησιμοποιούσαμε ε, ως ε, τροφή, ζωοτροφή για τους χείρους και τα πουλερικά. Ε, ξέραμε γιατί, τότε δεν ξέραμε για τα ολεύκομα και την προέλευσή του. Οι διοξίνες βέβαια, οι διοξίνες φοβίζουν αμέσως τον κόσμο και δεν είναι δυνατόν να είναι οι ε, τιμές ε, οι ανώτατες τιμές διαφορετικές από ό,τι σε άλλα γεωργικά προϊόντα τα οποία παράγονται σε χερσαία συστήματα ας πούμε, στην ξύρα. Ποια είναι τα όρια ε, επιβάρυνσης αυτά τα οποία ε, έχουν οριστεί στην Ευρώπη. Μας ενδιαφέρει επίσης για το γάδο, το σολομό, τη ρέγγα και την Σαρδελόρεγκα. Αυτά τα τέσσερα κυρίως ε, αυτά είναι που δίνουν το ψωμί στις χώρες της Βαλτικής. Αλλά επειδή έχω, και το, έχω εδώ το συνάδελφο Παλέσα δίπλα μου, ξέρει και εκείνος ε, που, ποιο είναι το πρόβλημα. Καμιά φορά ο έλεγχος της αλίας επί χρόνια δεν γινόταν σωστά και είχαμε πρόβλημα με, μεγάλο εμείς με τα γερμανικά αποθέματα. Ονόματα δεν λέμε, αλλά είναι γνωστό πότε συνέβη αυτό και γιατί. Ευτυχώς τα αποθέματα του γάδου βελτιώθηκαν λιγάκι και μπορούμε να μιλήσουμε για βιώσιμη αλληλεία. Είναι καλό αυτό. Αλλά είναι σημαντικός και ο έλεγχος, η εποπτεία στην αλληλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Λάσεν, τώρα έχετε το λόγο. Όπως βλέπετε υπάρχει μια σειρά σχολείων, ερωτήσεων και αντιδράσεων. Παρακαλώ να απαντήσετε. Um, ε, ευχαριστώ πολύ. Δεν φανταζόμουν ότι τα αποθέματα Ρέγκας και Σαρδελόρεγγας στη Βαλτική θα προκαλούσε τόσο ζωηρή συζήτηση και ενδιαφέρον. Αλλά ε, βεβαίως αντιλαμβάνομαι το λόγο. Για να δω τώρα αν θα μπορέσω να απαντήσω. Πρώτο σχόλιο. Όταν παράγει κανείς ηχθιάλευρα και ηχθιέλεα, αυτή είναι μία κατηγορία προϊόντος. Δεν είμαι ειδικό βέβαια, αλλά παίρνει κανείς νοπό ψάρι και κατόπιν επεξεργασίας παράγεται το ηχθιάλευρο και το ηχθιέλεο. Τώρα, έγινε μία ερώτηση σχετικά με τον παράγοντα μετατροπής. Δεν έχω τα στοιχεία, αλλά ασφαλώς μπορώ να ψάξω τα στοιχεία και να σας δώσω αργότερα. Χονδρικά, παίρνουμε το πρωτογενές υλικό, αφαιρείτε το νερό, ουσιαστικά κατά 70% της εκφόρτωσης. Άρα δηλαδή ως προς το 1 τρίτο, κατά το 1 τρίτο χρησιμοποιείται για την παραγωγή ηχθιαλεύρου και ηχθιαλέου. Το νερό είναι βασικό συστατικό βεβαίως για όλα τα ψάρια. Uh, in terms of the production, fish meal and Λοιπόν, ηχθιάλευρα και παράγονται στην Δανία. Ιδιαίτερος δηλαδή ε, δανέζικας και σουηδικά πλοία εκφορτώνουν στη Δανία το αλιεύμα που αλλιεύουν στην ανατολική πλευρά της θαλάσσης. Και στη Δανία υπάρχει ένα εργοστάσιο και οι πλειοκτήτες των σουηδικών ε, πλοίων κατά το παρελθόν υπήρχε και ένα εργοστάσιο στην Σουηδία αλλά ε, αυτό έκλεισε και οι Σουηδοί αγόρασαν ένα τμήμα του δανέζικου εργοστασίου στο Σκέν. Τώρα, Το πρόβλημα ότι δεν ξέρουμε ακριβώς τα στοιχεία είναι ότι δεν ξέρουμε ε, το, τη συνολική ποσότητα των εκφορτώσεων. Γίνεται δειγματοληψία. Η δειγματοληψία πριν από την 1η Ιανουαρίου δεν συνδεόταν με την παραγωγή, συνδεόταν με την εκφόρτωση του προϊόντος και μετά επιβεβαιώνεται αν πρόκειται για ρέγγα, ε, σαρδελόρεγγα ή οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό λοιπόν είναι δύσκολο να επανέλθει κανείς και να ε, μιλήσει για ακριβείς ποσότητες. Άρα λοιπόν έχουμε ακριβείς ε, αριθμούς για την ποσότητα της ρέγγας που έρχεται από διάφορες περιοχές της Βαλτικής, της Βόρειας Βαλτικής. Έχουμε πολύ ακριβή στοιχεία για το τι παράγει κάθε εργοστάσιο, αλλά αυτό, αλλά όμως δεν ξέραμε, δεν ξέραμε από πού προμηθεύεται την πρώτη ύλη το εργοστάσιο, αν δηλαδή την προμηθεύεται από τη Βόρεια Θάλασσα ή από κάπου αλλού. Μπορεί κανείς απλώς να εικάσει ως ένα βαθμό, αλλά δεν υπάρχουν ακριβείς αριθμοί, ακριβείς στοιχεία ως προς αυτό. Αυτό είναι ο για τον οποίο δεν μπορώ να σας πω ότι 297.522 τόνους, α πούμε, να σας πω ένα νούμερο συγκεκριμένο. Έγιναν πολλές ερωτήσεις σχετικά με την ε, ρέγγα της Δυτικής Βαλτικής. Αυτή η ρέγγα, αυτά τα αποθέματα έχουν κάποιο πρόβλημα τα τελευταία χρόνια, διότι η αναπαραγωγή γίνεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή που δεν μπορώ να προφέρω καλά. Ωστόσο, από αυτά, στα αυτά τα αποθέματα, από αυτά τα αποθέματα δεν υπάρχει βιομηχανική παραγωγή. Πρόκειται για μικρές ποσότητες ουσιαστικά που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανθρώπινη κατανάλωση και πηγαίνουν στη βιομηχανική αλεία. Αλλά η βιομηχανική αλεία δεν γίνεται σε αυτές τις περιοχές. Γι' αυτό το συμπέρασμά μου είναι ότι η βιομηχανική αλεία δεν επηρεάζει αυτά τα αποθέματα στη Δυτική Βαλτική. Ε, υπάρχουν ε, ενδεχομένως ε, άλλα λιεύματα που επηρεάζονται, άλλες ε, άλλα παραλιεύματα, αλλά όχι η ρέγγα. Γιατί αυτή η συγκεκριμένη ρέγγα έχει την κακή συνήθεια να αναπαράγεται στη Δυτική Βαλτική. Αλλά εμείς μιλάμε για την για τη Ρέγκα και τη Σαρντελόρεγκα που αναπαράγεται στην Ανατολική Βαλτική. Τώρα ερχόμαστε στη φιλανδική παραγωγή, η οποία και αυτή, τα φιλανδικά αλλιεύματα, που και αυτά προορίζονται για μηχανικούς σκοπούς. ουσιαστικά για, για υδατοκαλλιέργειες. Α, και παραγωγή γούνας επίσης. Δηλαδή χρησιμοποιείται για την εκτροφή αλεπούδων και τη μετέπειτα παραγωγή ε, γούνας. Το 50% ή ίσως και το 60-65% των εκφορτώσεων των Φιλανδών ε, πάει για αυτό το σκοπό. Τα στατιστικά στοιχεία έρχονται από το Φιλανδικό Ινστιτούτο και μπορείτε να βρείτε όλα τα στοιχεία στην ιστοσελίδα της, ε, του Ινστιτούτου αυτού. Αλλά πρόκειται αποκλειστικά για τα φιλανδικά στατιστικά στοιχεία. Τώρα, ηχθιάλευρα και ηχθιέλεα που χρησιμοποιούνται για την υδατοκαλλιέργεια ε, ουσιαστικά χρησιμοποιούνται στην Νορβηγία και την Σκοτία. Είναι ουσιαστικά οι δύο χώρες που παράγουν σολομό και χρησιμοποιούν τα ηχθιάλευρα και τα ηχθιέλεα. Χρειάζεται και λίγο υπάρχει ας πούμε μια μονάδα ε, στην Νορβηγία. Η Νορβηγία παράγει ένα εκατομμύριο τόνους ε, ε, ε, σολο, σολομού. Και επίσης... Και επίσης ε, χρησιμοποιείται για την παραγωγή πέστροφας. Έγινε αναφορά σε μελέτες σχετικά με την αναπαραγωγή. Παγκοσμίω θεωρείται βασικό πρόβλημα το γεγονός ότι η δατοκαλλιέργεια που ανθεί παγκοσμίω απαιτεί μεγάλες ποσότητες ηχθιαλεύρων και ηχθιελαίων. Γίνονται πάρα πολλές έρευνες γύρω από αυτό το ζήτημα. Χρειάζεται, χρειάζεται όμως αυτό για την, για την πρωτεΐνη. Ε, μπορεί κανείς ε, να ισχυριστεί ότι θα μπορούσε να, να χρησιμοποιηθούν άλλα είδη ντιλάπια και άλλα είδη. Αν θέλετε την προσωπική μου γνώμη ως προς τις προοπτικές, εγώ είμαι πάντα αισιόδοξο. Ξέρετε, πιστεύω απολύτως τους χημικούς. Η γυναίκα μου είναι χημικός και είμαι βέβαιος ότι μπορούν να τα φτιάξουν όλα. Όχι βεβαίως αύριο το πρωί ενδεχομένως, αλλά σε λίγα χρόνια είμαι βέβαιος ότι θα το κάνουν. Ε, αρκετές ερωτήσεις ε, αφορούσαν τον, ε, την όλη αλυσίδα του γάδου, ρέγγας κλπ. Οι μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει τέτοια σχέση πρέπει να δει κανείς αν θέλει να κάνει ε, μηχανική ε, οικοσυστημάτων. Απλώς τώρα εγώ λέω έτσι μια ιδέα ως παράδειγμα ε, οι σαρδελόρεγγες τρώνε γάδους και τα μοντέλα που έχουμε δείχνουν, τα πρότυπα δηλαδή, δείχνουν ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι σε αυτό το τομέα. Υπήρξε μια μελέτη η οποία ε, δημοσιεύθηκε από το ε, Συμβούλιο Υπουργών των Σκανδιναβικών ε, χωρών, που μια μελέτη η οποία με λεπτομερή τρόπο μελέτησε αυτά τα ζητήματα και κατά τη γνώμη μου πρόκειται για μια Ε, συζήτηση σε ποιο βαθμό θέλει κανείς να αναλάβει το ρίσκο ή όχι. Η δική μου. Η δική μου προσωπική αντίληψη είναι ότι τα πράγματα βαίνουν ομαλώς, εκτός και αν κάτι έκτακτο συμβεί. Αυτή είναι η δική μου προσωπική αντίληψη. Νομίζω ότι η Ζαμπέλα Λεβίν ρώτησε για ποιο λόγο δεν μπορούμε να ε, χρησιμοποιήσουμε σημεία αναφοράς βιομάζας και για τη Βαλτική και χρησιμοποιούμε μόνο ε, στοιχεία περιθνησιμότητας. Κοιτάξτε, προφανώς υπάρχει κάποια ποσότητα, πούμε. Δηλαδή ένας τόνος ε, γάδου για δέκα τόνους ρέγγας. Τούτο σημαίνει ότι μπορεί κανείς σε έναν βαθμό να λέει ότι η Βαλτική συνολικά μπορεί να προσφέρει αυτό που έχουμε ανάγκη. Το τι, το τι ακριβώς όμως μπορεί να προσφέρει είναι πολύ πιο δύσκολο να απαντηθεί. Τελευταίο σημείο. τιμές. Καλής ρέγγας. Μεγάλη ελέγγα δηλαδή. Πόσο υψηλότερη είναι η, ε, πόσο υψηλότερη είναι η τιμή μιας καλής ρέγγας σε σχέση με τη ρέγγα που θα γίνει χθιάλευρο ε, για να τα φάνε τα ψάρια ή οι αλεπούδες. Αν ε, γινόταν μια ανάλυση, ε, θα κατέληγε κανείς στο συμπέρασμα ότι το κόστος για την βιομηχανική αλία είναι πάρα πολύ χαμηλό. Δηλαδή απλώνει κανείς τα δίκτυα του και μαζεύει ό,τι βρει. Τα ψάρια για ανθρώπινη κατανάλωση έχουν διαφορετική δομή αλίευσης. Ε, τώρα, ως προς τα έσοδα τα... και συγκριτική μελέτη μεταξύ των δύο, δεν έχει γίνει. Ότι τουλάχιστον εγώ δεν έχω συγκριτικά στοιχεία και δεν είμαι οικονομολόγος για να σας τα πω. Then the Τελευταίο σημείο. Ε, έγιναν σχόλια σχετικά με τα δείγματα. Εγώ μπόρεσα να βγάλω 150 δείγματα για το 2010 και υπάρχουν αντίστοιχα ε, στοιχεία για το 9. Και από τη Δανία έχουμε στοιχεία για τις εκφορτώσεις ε, για βιομηχανική χρήση. και ε, ε, τα τελευταία χρόνια ξέρουμε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ως προς τα ηχθίδια ή τα νεογνά ψάρια ε, ρέγγας στη Βαλτική. Και λίγο πολύ τα στοιχεία είναι συγκρίσιμα ας πούμε με τη Βόρεια Θάλασσα. και ε, ως προς τη σύνθεση των ειδών νομίζω ότι η δειγματοληψία ή τα δείγματα μάλλον ήταν απολύτως επαρκή. And Τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς το γάδο. Μην ψάχνετε ψήλους τάχυρα. τα παραλιεύματα σε γάδος αυτές τις ε, περιοχές είναι πάρα πολύ χαμηλά, ελάχιστα. Πιστεύω λοιπόν ότι το επίπεδο δειγματοληψίας είναι πολύ καλύτερο εδώ σε σχέση με τη Βόρεια Θάλασσα, διότι η σύνθεση των ειδών είναι απλούστερη εδώ. Έχουμε απλώς ρέγγα, σαρδελόρεγγα και παρεμφερή. Έγιναν και διάφορα άλλα σχόλια για τον έλεγχο. Είναι εκτός της μελέτης όμως που εγώ σας παρουσιάζω. Και και υπήρξαν και κάποια σχόλια σχετικά με τις κλειστές περιοχές, κλειστοί, κλειστές λεκάνες αν θέλετε και ιδιαίτερα όσον αφορά τις ε, περιοχές αναπαραγωγής του γάδου. Ε, αυτά ενδεχομένως να είχαν κάποια αξία αν αναφερόμασταν στο γάδο, αλλά ε, στην περίπτωση της ε, Ρέγκας και Σαρδελόρεγκας δεν έχουν καμία σημασία. Δεν έχω άλλα σχόλια να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ερωτήσεις και για τα σχόλιά σας. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Λάρσεν. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θέλει κάποιος ο συνάδελφος το λόγο. Ε, τότε και πάλι ευχαριστούμε τον κύριο Λάση για την ε, εξαιρετική σας παρουσία. Και τώρα ολοκληρώσαμε το 18ο σημείο. Και επομένω πάμε στα διάφορα. Έχετε το λόγο κύριε Γκρόμπατσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω, ίσως ε, το, το, το, παρακάνω σήμερα όσον αφορά το πώς συχνά ζητώ το λόγο. Όμως, μιλήσαμε για την αντιπροσωπεία του Γκτάνσκ. Του Και θέλω σε σχέση με αυτό να προσθέσω ορισμένα πράγματα. Το ότι δηλαδή Είναι τελικά πολύ λεπτό αυτό το θέμα και επομένω θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και πότε θα υπάρξει ένα κείμενο και κάποια έκθεση. Πρώτα-πρώτα συμπαθούμε γιατί δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην αντιπροσωπεία. Έπρεπε να λύσω ένα πρόβλημα όσον αφορά τι πολωνικέ ακτέ. Όπου καταβάλλεται προσπάθεια να κλείσουν ορισμένα τμήματα του πανεπιστημίο που εκπαιδεύει ειδικού για την αλληλεία επιστήμονες. Και επομένως οι προσπάθειες μου είχαν στραφεί προς τα εκεί. Τώρα, ε, αυτή την επιχείρηση που θα πήγαινε την προσωπία μας. Εκεί τελικά δεν μπόρεσαν να πάνε δεν μπορούσαν να επισκεφθούν την επιχείρηση παρά το ότι ή στα έγγραφα αναφέρεται ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ασχοληθεί με την πρόθεση τέτοιων δραστηριοτήτων και αυτή η επιχείρηση είναι η κορυφαία, η πρωτοπόρωση σε αυτόν τον κλάδο. Και τώρα, λόγω της οικονομικής κρίσης, λόγω των ποσοστώσεων που έχουν επιβληθεί, λόγω την, αλλαγής όσον αφορά την ιδιοκτησία, θα ε, έχουμε 20 άτομα που θα χάσουν τη δουλειά τους και βέβαια είναι πάρα πολύ θυμωμένοι οι αλλοί Επίσης βέβαια διαδόθηκαν τα κακανέ πάρα πολύ γρήγορα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θέλησε να το συζητήσει. Οπότε εγώ θέλω, θέλω κάτι να να ζητήσω και κάτι να προτείνω. Θα ήθελα να καλέσουμε εδώ τους εργαζομένους σε αυτή την επιχείρηση. Να συναντήσουν την πρόεδρο. Αλλά και τους συναδέλφους. Όποιον ενδιαφέρεται. Όταν μπορούσαν να συμμετάσχω στα έξοδα για το ταξίδι αυτό, γιατί αποκομίστηκε πάρα πολύ άσχημη ε, απάντηση για το μέλλον. προκειμένου να συζητηθεί πολύ αυτό το θέμα και επομένω το πρόβλημα αυτό θα ξαναρθεί στην επικαιρότητα. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να σώσουμε τους ε, αλληλείς, να τους βοηθήσουμε για το μέλλον Και νομίζω ότι ήταν ντροπή που η αντιπροσωπή του το μόνο που ασχολήθηκε ήταν ξενάγησε στα μεσαιωνικά τείχη. Με την έκθεση να το συζητήσουμε. Να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βαρέσα. Μας εξήγησε ο Βαλέσα Εγώ πάντως δεν συμφωνώ ότι πήγαν και για βολτούλα, για εκστρομή οι βουλευτές. Αυτό σα το λέω ε, αμέσω τώρα πριν ξεκινήσουμε. Βαλέσα. Κύριε συνάδελφε, γιατί θα πρέπει να τα λέμε έτσι ανοιχτά μπροστά στην Επιτροπή για αυτή την σκούνερ. Κάτι να τα πούμε μεταξύ μας. Δηλαδή να πούμε ότι συναντήσαμε εκπροσώπους της Κούνερ. Αν θέλετε να βγάλετε τα άπλητά μας στη φόρα, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο. Ε, δεν είναι δυνατόν να λέτε ότι πήγαμε μόνο και μόνο για ξενάγηση στα μεσονικά τείχη. Ε, ε, επισκεφθήκαμε και μία αγορά, ψαραγορά, εκεί όπου διαμορφώνεται η πρώτη τιμή. Δεν είναι δυνατόν να μας ε, κατηγορεί κανείς ότι ε, δεν κάναμε το καθήκον μας. Και είναι πραγματικά ε, άστοχο αυτό το οποίο κάνατε το να μας προσβάλλει με αυτόν τον τρόπο. Μισό λεπτό, αν δεν σας πειράζει, να σας πω εγώ. Να μιλήσω εγώ γιατί δεν θέλω να τσακωθείτε. Ούτε με ενδιαφέρει, ούτε μ' αρέσει, ούτε συμφωνώ να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσατε εσείς να έρθετε, τι να κάνουμε. Τη μέρα που θα παρουσιαστεί η έκθεση, τότε μπορούμε να το συζητήσουμε. Άρα, θα δούμε τι θα γίνει στην επόμενη συνάντηση που έχουμε την παρουσίαση των πεπραγμένων στο ανακοινώσεις της ε, Προέδρου για τις αποφάσεις των συντονιστών. Όπου δεν υπάρχει ένσταση, θεωρώ ότι εγκρίνονται. Ημερομηνία τη προσεχού συνεδριάζω στι Βρυξέλλε. 15 Ιουνίου. 3 με 6,5 και 16 Ιουνίου. 9 με 12,5. Σα ευχαριστούμε. Πέρα συνεδριάζω.